of the Parliamentary last month. Περνάμε στο θέμα που είναι η η ανταλλαγή απόψεων με την ε, κυρία Γκαμπριέλα Μπαριών, που είναι πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Ένωση σχετικά με το ρόλο των βουλευτών στι οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά θέματα. Η IPU, η Διακοινοβουλευτική Ένωση, είναι πολύ σημαντική ε, για τη δουλειά των βουλευτών ανά τον κόσμο. Η πρόεδρος ε, της ε, Διακοινωνιστικής Ένωσης ε, συμμετείχε τους τελευταίους μήνες και σε διάφορες άλλες συζητήσεις, άρα δηλαδή βλέπουμε ότι έχετε την εμπειρία για το τι θα μπορούσε να επιφέρει αυτή η συνεργασία, ποια είναι τα ωφέλη που θα μπορούσε να φέρει στην κοινοβουλευτική διπλωματία. Βεβαίως ε, θα μπορούσα να φέρω πολλά πράγματα για σας και για την εμπειρία σας, αλλά ε, δεν θα προσθέσω τίποτα άλλο ε, και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λάγκε. Για μένα θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ. Ήμασταν μαζί στη Γενέβη, τώρα βρίσκομαι στην έντρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους σας. Και ε, θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω στα ισπανικά, γιατί έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συνεδριάσεις και έτσι έχω κουραστεί λιγάκι και ε, προτιμώ να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο οι κανόνες, οι προκλήσεις, οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα την οποία δεν θα φανταζόμουν ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Κάποια παραδείγματα και μοντέλα που θεωρήσαμε ότι θα υπάρχουν για πάντα σήμερα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαμε ότι το πολυμερές σύστημα, η παγκοσμιοποίηση, το εμπορικό άνοιγμα είναι οι θεμέλιες λύθη για οποιαδήποτε οικονομία. Σήμερα αντιθέτω βλέπουμε ότι σε ορισμένες ισχυρές οικονομίες του πλανήτη μας αυτές οι αξίες, αυτές οι αρχές, αυτή η αφήγηση τίθεται από αμφισβήτηση. Και γι' αυτό το λόγο η δουλειά των βουλευτών και η κοινοβουλευτική διπλωματία γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Και ε, βεβαίως ε, εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις στα παραδοσιακά πρότυπα διπλωματίας, όμως στην κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε την επικοινομορφία, την πολιτική, την, τον ιδεολογικό πλουραλισμό που εκπροσωπεί ολόκληρη την κοινωνία και η κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί γι' αυτό το λόγο να συνάψει δεσμούς με μεγαλύτερο βεληνικέ, μεγαλύτερη εμβέλεια και σε μεγαλύτερο βάθο χρόνου. Ε, τις νέες προκλήσει φαινόταν στο παρελθόν θα αντιμετωπίζουν μόνο οι κυβερνήσει. μάλιστα οι κυβερνήσεις που δεν έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο περιθώριο. Ωστόσο σήμερα βλέπουμε επιβολή δασμών, βλέπουμε εμπορικούς πολέμους και αυτός είναι μηχανισμός πολιτικών ανταλλαγών. Δηλαδή αυστηρά οικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται σήμερα από κυβερνήσεις για διάλογο ή κυρίως για πολιτική αντιπαράθεση. Και εκεί έγκυται και το πρόβλημα το ευρύτερο του πώς κανείς προσεγγίζει τις συζητήσεις με εθνικιστές που υιοθετούν εθνικιστική αφήγηση π.χ. ή διάφορα άλλα θέματα. Προς τα πού οδεύει ο κόσμος μας, τι θα πρέπει να περιμένουμε σε 10 χρόνια από σήμερα. Εάν θέσουμε το ερώτημα αυτό, πολύ δύσκολα θα δώσουμε απαντήσεις. Κάποιες μελέτες μας λένε σήμερα ότι αναλόγως με τις τεχνολογικές εξελίξεις, πολλά επαγγέλματα που γνωρίζουμε σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν πια. Όμως αυτά που θα δημιουργηθούν τα επόμενα 10 χρόνια είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν αδύνατο να τα αντιληφθεί και να τα συλλάβει κανείς διανοητικά. Τώρα, ποιε θα είναι οι ευκαιρίε για του νέου από πλευρά κοινωνική ασφάλισης, από πλευρά συνταξιοδότηση σε 10 χρόνια από τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να δοθούν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί στην οικονομία και το πώ θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια. Τι περιμένει κανεί από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση. Καταρχά πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική πολιτική μα ατζέντα. Έχουμε Επιτροπή για την Αηφόρο Ανάπτυξη στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και θέλουμε να διευρύνουμε την εντολή εντολή αυτή τη Επιτροπή και να την κάνουμε ακόμα και πιο εξειδικευμένη. Μπορεί όμω αυτό να χρειαστεί χρόνο για να γίνει. Και όπω είπε και ο πρόεδρο Μπερτ Λάγκε, έχουμε τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη στο πλαίσιο του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και θα πρέπει να δώσουμε, να εμφυσίσουμε νέο περιεχόμενο στο θεσμικό αυτό όργανο, ώστε να καταλήξει σε μεγαλύτερε προτάσει. Είναι μεγάλη ευθύνη την οποία μοιράζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση. Δηλαδή, να είμαστε υπέρμαχοι της πολυμερούς προσέγγισης μέσα από σαφείς κανόνες και θέσεις που αναδεικνύουν και καταδεικνύουν ότι ο καλύτερος τρόπος να υπερασπιστεί κανείς την πολυμερή προσέγγιση είναι να δείξει τα αποτελέσματα και το περιεχόμενο και την ουσία του. Και έχουμε ένα νέο μηχανισμό τη συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών, των χωρών G20 και αυτό το ονομάζουμε P20, Parliament 20 δηλαδή. Και αυτό, που, αυτό το σχήμα δεν έχει συγκεκριμένους κανόνες και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Έτσι έχουμε πολύ σημαντικές συζητήσεις που πολλά υποσχόμενες, κάποιες άλλες αφήνουν ζητήματα εκρεμή. Σε κάθε περίπτωση ένας μηχανισμός είναι αυτός ο οποίος προχωρά και μάλιστα με βήματα αποφασιστικά. Ο μηχανισμός της διάσκεψης των προέδρων των κοινοβουλίων των χωρών του G20, το P20 δηλαδή. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποκριθούμε στις προκλήσεις του σήμερα και να προβλέψουμε αυτό που θα συμβεί και στο μέλλον. Και ε, δεν χρειάζεται να είναι κανεί μάντη για να μαντέψει ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, θα έχουμε οικονομική επιβράδυνση τα επόμενα χρόνια. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είναι σαφέ. Είναι πολύ σαφέ ότι ο κόσμο δεν έχει ανακάμψει πλήρω από τη χρηματοπιστωτική και χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Είναι προφανέ ότι η αντιπαράθεση μεγάλων ε, οικονομικών δυνάμεων, υπερδυνάμεων, θα συνεχιστεί μέσα από ένα μηχανισμό που θα συγχαίει το πολιτικό σκέλο με το οικονομικό. Αυτά είναι προφανή και σαφή. Ωστόσο, άλλε χώρε που δεν το φανταζόμασταν αρχίζουν να προσχωρούν στο ελεύθερο εμπόριο. Άλλα συστήματα, άλλα προγράμματα με πολυμερή προσέγγιση δεν κατάφεραν να λύσουν πολύ περίπλοκα προβλήματα. Εμείς ως βουλευτές, εσείς ως βουλευτές έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη. Καταρχάς εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας. Εμείς ε, συντάσσουμε προϋπολογισμούς, ε, ε, παρακολουθούμε και ελέγχουμε το κυβερνητικό έργο. Και άρα εμείς που ασχολούμαστε με την πολυμερή προσέγγιση πρέπει να επιστρέφουμε στις πατρίδες μας με λύσεις και απαντήσεις αφέστατες. Εάν σήμερα μας θέσουν την εξής ερώτηση, ο καθένας στη χώρα του, τι θέσεις έχουμε για την απασχόληση των νέων για τα επόμενα 20 χρόνια, πρέπει να ξέρουμε τι θα απαντήσουμε να ξέρουμε τι μας ρωτούν οι νέοι, ε, ποιες είναι οι ελπίδες που μπορούν να τρέφουν για το κατά πόσο θα έχουν κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη, να ξέρουμε τι θα απαντήσουμε, πώς θα μας εγγυηθείτε ότι θα υπάρχει ίσως μισθός μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίση απασχόληση, για ίδια απασχόληση. Πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Αυτή η πολιτική και η οικονομική ατζέντα λοιπόν μας αφορά. Και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας προσκαλέσω, Πρόεδρε, στην επόμενη συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης τον επόμενο Απρίλιο του 2020. 2020. Βασικό αντικείμενο θα είναι η οικονομική ατζέντα, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε απαντήσεις για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη μας, τα οποία είναι δυσεπίλητα. Και επιμένω επίσης, γιατί είναι και απότοκος της κρίσης του 2008 αυτό, ε, είμαστε μάρτυρες μιας νέας αδράνειας ε, τα τελευταία χρόνια που θα οξυνθεί. Αυτά καταρχάς. Άλλα θέματα που θεωρούμε σημαντικά είναι η ενίσχυση της κοινοβουλευτική συνεργασίας. Μεταξύ των βουλευτών θα πρέπει να υπάρχει διπλωματία, να μην έχουμε μόνο διάλογο, ψηφίσματα και δηλώσεις και εκθέσεις, αλλά να έχουμε και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ένα από τα θέματα που θα μπορούσαμε να ε, το δουλέψουμε από κοινού είναι το εξή. Πώς οι χώρες και τα κοινοβούλια που ήδη ε, έχουμε σημαντική εμπειρία από πλευράς εμπορίου, από πλευράς επενδύσεων, συνθήκων, συμβάσεων, πώς μπορούμε αυτές τις εμπειρίες να τις ε, συγχωνεύσουμε, να τις συγκεράσουμε και να τις μοιραστούμε με τις περιοχές και περιφέρειες που κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα σε αυτό το τομέα. Να μιλήσουμε και για τα καλά και για τα κακά δηλαδή όλων αυτών των συμφώνων φωνιών. Εγώ είμαι από το Μεξικό. Έχουμε 25 χρόνια πολιτική ελευθέρου εμπορίου στο Μεξικό με διάφορα λάθη. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη εμπειρία. Η Χιλή έχει το μεγαλύτερο αριθμό συμβάσεων ελευθέρου εμπορίου με άλλες μετρήτες χώρες. Έχουμε εμπειρία τεράστια στην επιμελητία, στα logistics, στον εφοδιασμό στη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη δηλαδή έχει. Άρα αλλά άρα θα μπορούσαμε να ε, συγκεράσουμε αυτές τις απόψεις για να μάθουμε ένας από τον άλλον και να καταλήξουμε στην ουσία. Να έχουμε λοιπόν ανταλλαγή γνώσεων όπου όλοι θα πλουτίσουν τις γνώσεις τους. Και νομίζω ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει πολύ, πολλά να προσφέρει σε αυτό το επίπεδο. Πώς θα βοηθήσει ο ένας τον άλλον, πώς η αλληλεγγύη μεταξύ ημών θα μεταφραστεί σε βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τους οποίους εκπροσωπούμε. Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, που πιστεύω ότι είναι και δικό σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία διάσταση σε όλες τις διαδικασίες, μεγαλύτερη λογοδοσία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό είναι μέρος της εντολής που έχουμε στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και θέλουμε όλες αυτές τις διαδικασίες να τις εξετάζουμε εκ του σύνεγγυς μαζί με τον ΠΟΕ, με τα Ηνωμένα Έθνη και με αυτό το θεσμικό όργανο του P20, των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών ε, των, ε, του G20. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ε, για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Στον κύριο Χάνσεν, εκ μέρους του ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στη δική σας τη γλώσσα τότε και εγώ. Θα ήταν σημαντικό για μένα να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο και από κοινού για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών με το Μεξικό αλλά και με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ε, υπάρχει συμφωνία με το Ιμερικοσούρ που ε, προσεχώς ε, θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο και πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε βιώσιμες λύσεις. Παραδείγματο χάρη για το πρόβλημα των ε, πυρκαγιών στην περιοχή του Αμαζονίου και άλλα. Υπάρχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά εδώ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία ώστε και άλλη πλευρά να ε, βοηθήσει για να μπορέσουμε να διαφωτίσουμε περισσότερο τα πράγματα και να βρούμε λύσεις και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Με εντυπωσιάσατε. Κάθλιν Φαν Σοσιαλιστές και Δημοκράτης. Ε, μακάρι να μπορούσα και εγώ να μιλήσω ισπανικά. Ε, προσπαθώ να μάθω λίγο Ισπανικά, γιατί είναι γλώσσα που μιλάτε σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα μιλήσω όμως Αγγλικά, την άλλη γλώσσα που μιλάνε όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει συνεργασία για θέματα εμπορίου. Ε, Έχω δύο θέματα και δύο ερωτήσεις. Δύο θέματα που θέλω να θίξω και δύο ερωτήσεις. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αγορά εργασία σε σχέση με τη βιωσιμότητα, οικονομικής φύσεως θέματα. Νομίζω όμως ότι λίγο πολύ εμφανίζεται και μία κρίση για την ίδια τη δημοκρατία και κυρίως για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό. Να το συζητήσουμε το Κοινοβούλιο και η IPU, η Διακοινοβουλευτική Ένωση. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα πολύ σημαντικό χώρο της δημοκρατίας, προάσπισης ε, ευρωπαϊκών αξιών, κράτους δικαίου, αλλά και στη μία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε προβλήματα για το κράτος δικαίου. Φύσατε πίεση στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Και θα ήθελα να γνωρίζω πώς εσείς αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα θέματα και πώς μπορούμε μέσω στενής συνεργασίας να τα αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού. Το δεύτερο που θέλω να θίξω είναι η βιωσιμότητα. Σήμερα το πρωί είχαμε μία μακρά συζήτηση για την Συμφωνία Εμπορικών Ανταλλαγών ε, με το Βιετνάμ. Θα συζητήσουμε και για συμφωνία με το Μερκοσούρ. Είναι ένα θέμα που πραγματικά βρίσκεται στην καρδιά των συζητήσεων στο Κοινοβούλιο. Το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό. Το εμπόριο από μόνο του είναι μια πολύ σημαντική αξία, αλλά πρέπει ε, να έχουμε τη διασύνδεση με τη βιωσιμότητα γνωρίζω τις χώρες ε, Μερκοσούρ και θα ήθελα να μας πείτε ε, ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με αυτά που ε, διαδραματίζονται στη Βραζιλία. Εκ μέρους της Renew είναι η πρώην φιλελεύθερη και νυν φιλελεύθερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Κάλσπρουρτ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Ε, πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Νομίζω ότι η εμπορική πολιτική είναι ένας τρόπος για να διαμορφώνεται, για να διαμορφωθεί η παγκοσμιοποίηση σε μια δύσκολη εποχή. Εμείς πιστεύουμε στο εμπόριο, πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι κάτι καλό για την ανάπτυξη, την ευημερία και επίση ε, είναι πολύ καλό και για τις ανθρώπινες ε, σχέσεις. Νομίζω ότι φέρουμε όμως και κάποια ευθύνη. Ευθύνη να βρούμε τους ε, βέλτιστους κανόνες για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τις εμπορικές πολιτικές και τις εμπορικές συμφωνίες. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι το εμπόριο ε, πρέπει να γίνεται με βάση κάποιους ε, κανόνες ε, και κάποιες αρμοδιότητες. Όσον αφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, την ενσωμάτωση της εμπορικής πολιτικής στην παγκόσμια κλιματική πολιτική. Αυτό είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, όπως είπαμε και σήμερα το πρωί, ε, υπάρχει η δημοκρατία, υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και πρέπει να κάνουμε μία επιλογή. Πιστεύουμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, μπορούν να αποτελούν μία πλατφόρμα για να προαχθούν η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή πιστεύουμε ότι χωρίς συμφωνίες τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται συζητήσεις στα κοινοβούλια από ερετούς εκπροσώπους των πολιτών να συμπεριλαμβάνονται στις συζητήσεις αυτές πολύ άμεσα ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο αυτοί ε, που συμμετέχουν στις συζητήσεις ε, για την παγκοσμιοποίηση και τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά αφορούν τη ζωή μας, το περιβάλλον και αφορούν και στο μέλλον του πλανήτη. Με μεγάλη μου λοιπόν χαρά να ακούσω τις ε, απαντήσεις σε, όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν σήμερα επιτάπητος. Ε, ο κύριος Μπουρζουά είναι από το κόμμα των συντηρητικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία ε, πρόεδρος ε, της IPU. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, εμπεριστατωμένη εισήγησή σα ε, στον πέμπτο στόχο σας αναφερθήκατε στον διακοινοβουλευτικό διάλογο στην προαγωγή της εργασίας. Επισημάνατε ότι αλλάζουν οι καιροί, ότι υπάρχουν ε, ε, μεγάλες γεωπολιτικές μετατοπίσεις, εμπορικές συγκρούσεις που θα μπορούσαν να καταλήξουν και σε εμπορικούς πολέμους. Ε, παρουσιάσατε λοιπόν μια θέση και αυτό λιγάκι με εξέπληξε ότι ο διακοινοβουλευτικός διάλογος μπορεί να είναι ε, ένας ε, δρόμος ε, για να πλησιάσει μία πλευρά την άλλη. Και ρωτώ πώς ακριβώς το εννοείται αυτό συγκεκριμένα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μέσα από τον διακοινοβουλευτικό διάλογο. Και δεύτερον, πιστεύετε ότι όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχω κατά αυτά που είπε ο ο προτινόμενος επίτροπος κύριος Χόγκαν, ο οποίος ε, τάχθηκε υπέρ του ε, ευρωατλαντικού διαλόγου. Πιστεύετε κι εσείς ότι ο διάλογος ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Αμερικανικό Κογκρέσο ε, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να πλησιάσει η μία πλευρά την άλλη περισσότερο. Ο κύριος Σόλτς από την ΚΟΕ που είναι το αριστερό κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ε, παρατηρήσεις σας, τις αρχικές. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όλα αυτά που είπατε. Δηλαδή ότι ναι, μεν είμαστε η Επιτροπή Εμπορίου, αλλά γενικά πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην πραγματικότητα που επικρατεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε το θέμα από την προοπτική του διεθνούς εμπορίου, πράγματι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας ε, και για να μπορέσουμε τα επόμενα δέκα χρόνια να επιτύχουμε το θεματολόγιο των ΗΕ για το 2030. Αυτό, όλα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, άρα να αλλάξουμε κανόνες και να περάσουμε στην πραγματικότητα των οικονομιών. Να αναζητήσουμε ε, τα αίτια που οδήγησαν στην έκθεση της ΑΝΚΤΑΤ, προτάσεις δηλαδή για μια νέα παγκόσμια πράσινη συμφωνία. Ε, οι αρχές της Γενέβης το αναφέρουν αυτό, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να ε, αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Και εδώ ε, φτάνω σε ένα από τα ερωτήματα, το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανασυνδέσουμε τις ε, δραστηριότητες των ε, κυβερνήσεών μας, ας πούμε του ΠΟΕ, σε κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Και οι εντολές ε, για διαπραγματεύσεις ε, θα πρέπει να δίδονται μόνο αφού προηγηθούν σοβαρές συζητήσεις για τους στόχους των διαπραγματεύσεων, για τις υποχρεώσεις. Νομίζω αυτό μπορεί να συμβάλλει στο να ε, συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι καλύτερα το τι ακριβώς κάνουμε σε διάφορους οργανισμούς. Και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω για όλα αυτά τα θέματα. Και τελευταίος ο μιλητής είναι ο αντιπρόεδρος ε, του ε, κοινοβουλίου μας, ε, ο κύριος Πέντρος Σίλβα Περέιρα. ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ στη δική μου γλώσσα, όπως έκανε και η προσκεκλημένη μας. Θα μιλήσω εγώ πορτογαλικά. Μοιάζουν πολύ άλλωστε με τα ισπανικά. Ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω την ε, Κοινοβουλευτική Ένωση γιατί έχει μπει ως θέμα ε, ενός συνεδρίου στο οποίο αυτή τη στιγμή τον δυτικό έχει η Ιαπωνία, στο ότι θα αποφασίσει, τα θέματα βιώσιμου εμπορίου. Είναι μεγάλη προτεραιότητα στη συνεδρίαση αυτή το θέμα του δικαιομπορίου. Υπάρχουν επίμαχα σημεία με τις διάφορες εμπορικές συμφωνίες. Για να τα αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να εστιάσουμε στο περιεχόμενο. Δεν είναι θέμα διαδικασίας τύπου, αλλά περιεχομένου, ουσίας. Οι εμπορικές συμφωνίες, κατά την άποψή μας, θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, και σε επιταγές ε, της πραγματικότητας και των νέων γενεών. Άρα έχουμε τα κεφάλαια της βιώσιμης ανάπτυξης πλέον που πρέπει να περιλαμβάνονται και αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Σίγουρα βέβαια και στα διαδικαστικά πρέπει να δώσουμε σημασία, αλλά κυρίως στην ουσία που είναι τα περιβαλλοντικά κοινωνικά ζητήματα που απαιτούν απάντηση μέσω των εμπορικών συμφωνιών. Αλλιώς δεν θα αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά και αποφασιστικά το πρόβλημα. Σίγουρα χρειάζονται διαδικασίες που θα εγγυώνται τη διαφάνεια των διαδικασιών. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολύ θετική εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολύ σημαντικά βήματα καλύτερη δημοσιοποίηση και προβολή των ζητημάτων και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Για συμμετοχή του Κοινοβουλίου, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών και τις αλλαγές που αυτές συνεπάγονται. Πρέπει να δούμε επίσης και τη διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου της πρακτικής εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών. Δεν μιλάω για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών, αλλά για την εφαρμογή πλέον των εμπορικών συμφωνιών. Τα Μάλλον τα κοινοβούλια πρέπει και αυτά να συμμετέχουν. Είναι σημαντικό. Και αυτό ε, να συμμετέχουν σε ισότιμο επίπεδο και με την κοινότητα των πολιτών. Άρα εδώ συμφωνούμε. Είναι κοινέ οι ανησυχίες μας και μπορούμε να συνεργαστούμε. Πρόεδρος, ήρθαν δύο καστερμένα αιτήματα. Ε, θα δώσω το λόγο για ένα λεπτάκι, καταρχάς τον κύριο Βίνκλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, που για το λεπτάκι που μου δίνετε, δεν θα το υπερβώ. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας κυρία Πρόεδρε της Δεκοινοβουλευτικής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία ε, και έχει όλο και μεγαλύτερο ε, λόγο. θα ε, νομίζω, και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις νέες μας εξουσίες. Το εμπόριο είναι μια αρμοδιότητα που έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συγκεκριμένα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπόριου είναι η καθήλυνα αρμόδια και στην κοινοβουλευτική διάσταση του ΟΗΕ και του ΠΟΕ συγγνώμη, και άλλων ε, φορέων ε, συμμετέχουμε και μπορούμε να επηρεάσουμε. Τι άλλη συνεργασία θα μπορούσαμε να έχουμε με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση σε θέματα εμπορίου κυρίως και βιώσιμης ανάπτυξης. Και η κυρία Ραφαήλ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση Στη σελίδα 21 στρατηγική σας για την περίοδο 17-21 λέτε ότι θέλετε να συμμετέχουν τα κοινοβούλια στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη. Τι έχετε κάνει για τη στρατηγική και το μέτωπο αυτό συγκεκριμένα. Με τα κοινοβούλια πώς θα συνεργαστείτε για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξης και σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο. Και δεύτερο, σελίδα 24 τη στρατηγική σας για την περίοδο 17-21 Πολύ σωστά λέτε ότι το εμπόριο είναι μοχλός τη παγκοσμιοποίησης. Μπορεί να βοηθήσει μια αλληλέγγυα βιώσιμη ανάπτυξη. Ποιο είναι ο ρόλο τη ένωση τη Δεκοινοβουλευτική, για την πρόθεση αυτή τη προσέγγιση. Ο Γκαμπριέλα. Γκαμπριέλα, ε, κάποιες λίγες μικρές ερωτήσεις. Να σας δώσω 9 λεπτάκια. Μια ώρα θα ήταν καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα κάνω ό,τι μπορώ να τα πω γρήγορα γρήγορα, αλλά δεν ήταν εύκολες οι ερωτήσεις. Είμαι Μεξικανή. Και είμαι μέλος ε, της ε, κοινοβουλευτικής ε, αυτής αντιπροσωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού και έχω συμμετάσχει και στο Eurolat ότι υπάρχουν καλοί μηχανισμοί κοινοβουλευτής δημοκρατίας, το ξέρω και λειτουργούν και σωστά. Πολύ καλά. Η η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού τα τελευταία, την τελευταία φορά που θυμάμαι ήταν πριν τρία χρόνια πριν να λάβω καθήκοντας πρόεδρος της ε, IPU. Ήταν μια καλή εμπειρία γιατί υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχει σίγουρα καλή παρακολούθηση, διαφάνεια, πολύ καλές διαδικασίες. Οπότε μπορείτε να μάθετε και πώς δεν πραγματεύονται οι αρχές σας τέτοιου είδους συμφωνίες. Αλλά εμείς δεν είμαστε ένα ισχυρό ε, κοινοβούλιο, είμαστε ένας κογκρέσου. Εσείς έχετε δυνατότητες επαφής και αλληλεπίδραση με τις αρχές. Όταν λοιπόν έχετε αυτές τις δυνατότητες διαλόγου, το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσεις εκφράζουν την πλειοψηφία και όχι την πολυμορφία, τον πλουραλισμό. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία όμως εκφράζει το λαό, τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι το εμπόριο είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι όμως ε, αυτός σκοπός. Είναι μέσο. Πριν από δύο-τρει δεκαετίε, ίσω πολλέ κυβερνήσει πίστευαν ότι το εμπόριο ήταν αυτό σκοπό. Ήταν ένα μαγικό εργαλείο, ένα μαγικό ραβδί. Αυτό είναι ένα σφάλμα. Και στο Μεξικό. Που πιστεύαμε ειλικρινά στο ελεύθερο εμπόριο. Και πιστεύω εγώ στο ελεύθερο εμπόριο. Δεν είναι όμω αυτή η μόνη απάντηση. Ο διάβολο, λένε, κρύβεται στι λεπτομέρειε. Και όταν μιλάμε για το εμπόριο, ναι, πιστέψτε με, κρύβεται εκεί μέσα πράγματι Σίγουρα με τις συμφωνίες μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, ε, ανάπτυξη των βιομηχανιών κτλ. Αλλά δεν υπάρχει βιομηχανικό σχεδιασμός. Αν δεν υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη ή μια σαφή στρατηγική ώστε τα διάφορα τμήματα, οι διάφορες περιοχές, περιφέρειες να υποφεληθούν των νέων εμπορικών ευκαιριών. Ναι, κάποιο μέρος της χώρας θα αναπτυχθεί, όπως σημαίνει με το κεντρικό ή βόρειο Μεξικό, αλλά το νότιο μέρος δεν επωφελείται. Και βέβαια μπορεί κάθε λεπτό να έχουμε συναλλαγέ ε, τη τάξη του ενό εκατομμυρίου δολαρίων με τη ΣΥΠΑ. Δεν πάνε όμω στον Νότο τα λεφτά αυτά. Ναι, μεν λοιπόν καλό και άγιο το εμπόριο, αλλά εξαρτάται από το πώ γίνονται ματεύσει και πώ εφαρμόζονται τα συμπεφωνημένα. Κύριε Λάγκε, ακούστε με. Εμείς θέλουμε φυσικά να συνεργαστούμε μαζί σας. Είναι πολύ καλή αυτή η συνεργασία μας και στο πλαίσιο του ΠΟΕΤΑ, πάμε και στη Γενέβη και πιστεύω ότι έχουμε τεράστιο δυναμικό και Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε πιο ενδιαφέροντα στήματα. Έχουμε εμπορικούς πολέμους, δασμούς και πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Και δεν μιλάμε μόνο για τον ΠΟΕ και τι γίνεται εκεί. Υπάρχει ο μηχανισμό παρακολούθηση τι γίνεται στον ΠΟΕ, ναι, αυτό το φόρμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και να ασχοληθούμε με το εμπόριο συνολικότερα. Υπάρχουν και άλλοι τομείς βέβαια συνεργασίας. Και επειδή υπόθηκε αυτό, Υπάρχει και ομάδα των 20, των G20, ευχαριστώ τον Πέτρο, και κάτι που μπορούμε να κάνουμε για την Αφρική, ίσως, με τις ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Να μην κάνουν τα λάθη που κάναμε πριν 25 χρόνια. Τον Απρίλιο συνεδριάζουμε, η συνέλευσή μας. Έχουμε εστιάσει σε οικονομικά θέματα, βέβαια, αλλά καλό να έρθετε όχι μόνο εσείς, Πρόεδρε, αλλά και άλλα μέλη τη επιτροπή σα η συνάντηση αυτή στη Γενέβη και αν έχετε άλλε ιδέε. Ευχαριστώ. Ό,τι μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μα είναι θετικό. Για τη δημοκρατία δεν μίλησα. Τα είπα σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θα κόψω λίγα αυτά που θέλω να πω. Ε, έχουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά υπάρχουν και άλλου είδου δημοκρατίε. Προεδρική δημοκρατία. Δεν είναι όλε οι χώρε κοινοβουλευτικέ δημοκρατίε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η νομοθετική εξουσία είναι στο επίκεντρο. Αν δεν έχουμε αντιπροσωπευτικά ισχυρά κοινοβούλια, ε, εκλεγμένα κοινοβούλια, δεν θα έχουμε ισχυρή δημοκρατία. Το μεγαλύτερο σφάλμα της γενιάς μας ήταν ότι τη δημοκρατία και ιδίως τη δημοκρατία ανθρώπινα δικαιώματα θεωρήσαμε δεδομένο. Ίσως να ήταν αυτό το μεγαλύτερο σφάλμα του αιώνα. Γιατί υπάρχουν αυταρχικά αλλά και λαϊκιστικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν αυτή την έλλειψη πάθους για τη δημοκρατία και τώρα ξαφνικά βλέπουμε αποτελεσματικέ κυβερνήσεις να είναι αυτές που είναι οι πιο αυταρχικές και που δεν σέβονται τα άνθρωπα δικαιώματα. Πρέπει να τους δείξουμε ότι δεν υπάρχει αντιστάθμιση μεταξύ δημοκρατίας και αποδοτικότητας. Δεν θα είναι εύκολο γιατί οι δημοκρατίες είναι προσιλωμένες στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τι πιστεύω ότι χρειάζεται. Πολιτική ηγεσία. Αλλά τη φοβόμαστε την πολιτική ηγεσία. Είμαστε σε μια χρονική στιγμή που ίσως έχουμε εντονότερες συζητήσεις και γίνονται πιο μεγαλόστομες δηλώσεις πριν από 15 χρόνια. Ε, εμείς οι βουλευτές δεν πρέπει να φοβόμαστε τη συζήτηση, το διάλογο, αντίθετα. Πρέπει να μας συναρπάζει αυτή η δυνατότητα και εδώ στα κοινοβούλια μπορούμε να βρούμε κοινό έδαφος και να καταλήξουμε σε κοινέ λύσεις. Αυτό είναι το καλύτερο με τον κοινοβουλευτισμό. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ε, σχολές σκέψης, αλλά ε, πέραν ε, του τρόπου σκέψης υπάρχει και ο τρόπος του να νιώθει κανείς στο μυαλό και η καρδιά πάνε μαζί και έτσι μπορούμε να κάνουμε αλλαγέ. Έχω επισκεφθεί όλο τον κόσμο. Ε, το ζήτημα τη πολιτικής ηγεσία το βλέπουμε παντού. Δεν αρκεί η νομοθεσία να είναι καλή. Πρέπει να φτάσουμε στην εφαρμογή. Μερκοσούρ και περιοχή Αμαζονίου, ναι, είναι πολύπλοκο όλη η περιοχή ε, καθίσατε πιο πολύπλοκε δυστυχώ. Όλοι έχουμε αντιμετώπιση προκλήσεις με την κλιματική αλλαγή. Δείτε τι γίνεται σε σχέση με την ανάπτυξη, με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Σε κάθε περιοχή. Πριν από δύο εβδομάδες έπρεπε να κάνω μια σχετική ομιλία. Η Ευρώπη δεν τα πάει και τόσο καλά σε ό,τι αφορά τα ωκεανούς, καλύτερα πρότυπα κατανάλωσης, ε, και υπάρχει και ένα άλλο, δεν το θυμάμαι, αλλά έχετε προκλήσει να αντιμετωπίσετε κι εσείς. Με βάση ένα σοβαρό site το οποίο συμβουλεύτηκα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το κατεπήγον του συστήματο. Ακούγονται φωνέ που λένε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια και τόσο σημαντική. Αρκεί να δει κανεί τι γίνεται στον πλανήτη. Δεν χρειάζεται να κάνει επιστήμονα, αρκεί ο κοινό νου. Αυτό που πιστεύω και επιτρέψτε να το πω μάθαμε στο Μεξικό ότι χρειάζεται μια νέα γενιά συμφωνιών και η Συμμαχία του Ειρηνικού ήταν ένας νέος τρόπος να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, όχι μόνο λόγω του εμπορίου, υπήρχαν και πολλές άλλες συνιστώσεις και δεσμεύσεις σε κλιματική αλλαγή και σε άλλους τομείς ε, ανήλυφθησαν δεσμεύσεις. Ναι, το εμπόριο, επαναλαμβάνω, είναι μόνο ένα μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πάρα πολύ γρήγορα μην άγχεστε, λέει ο πρόεδρο. Α, ωραία. Λοιπόν, δεικνοβουλευτικό διάλογο. Και εδώ δεν είναι αυτό ο σκοπό. Είναι όμω ένα ισχυρό εργαλείο. Παραδείγματο χάρη. Αν στενομένα Έθνη πάμε και προσπαθήσουμε να, βάλουμε, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι δύο χώρε που ποτέ δεν πρόκειται να μιλήσει μια στην άλλη. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό λόγω ε, του ότι είναι μια πολιτική δήλωση. Ε, είναι συμβολικά ε, σημαντική η πολιτική αυτή κίνηση και δεν θα την κάνουν, ακόμα και αν ήθελαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Εδώ υπάρχει πολιτική πολυμορφία και εκπροσωπούνται διάφορες θρησκευτικέ ομάδες κτλ. Ο διάλογος είναι διαφορετικός εδώ. Η δική μου εμπειρία, γιατί είχα πολλές συναντήσεις ε, με βουλευτές, κοινοβούλια, ε, για θέματα για τα οποία στη χώρα μου δεν έχουμε καμία συμφωνία ή καμία συνάντηση κτλ. Η εμπειρία λοιπόν της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι ότι πρώτον αποκομίζεις γνώση. Αν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ένα τον άλλο λίγο περισσότερο, μπορεί να βελτιωθεί πολύ πολιτική η ενσυναίσθηση υποτιμάται. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε αυτό. Η βάση της πολιτικής είναι γνώση. Και αυτός ο πλουραλισμός, αυτή η πολυμορφία είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ίσα ίσα είναι αυτό που κάνει τόσο σημαντικά τα κοινοβούλια ε, τα κάνει να είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας. Ε, και σίγουρα ο κοινοβουλευτικό διάλογος μπορεί να αποφορτήσει εντάσεις, έτσι έχει δείξει δική μου εμπειρία στην IPU. Κάποιες φορές ε, το πάθος δεν εύκολο να το αντιμετωπίσει κανείς, τα πάθη, αλλά πάλι με την πολυμορφία, τον πλουραλισμό μπορείς να βρεις λύση για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε πολλούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε πρωταθλητές στην IPU για την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση, UNDP λοιπά. Για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και βοηθούμε τα εθνικά κοινοβούλια να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν τους στόχους αυτούς. Πρέπει να κάνουν πολλά ακόμη. Μόνο το 10% των κοινοβουλίων ασχολούνται ενεργά με την επίτευξη αυτών των στόχων. Είναι πολύ περίεργο. Θεωρούν ότι είναι στόχος ε, και καθήκον της κυβέρνησης όταν μιλάμε για ένταξη, λέμε ότι πρέπει να μελετήσουμε την νομοθεσία σημαντικά, γιατί υπάρχουν, ε, συνολικά, γιατί πολλά νομοθετήματα περιλαμβάνουν διακριτικέ διατάξει, ιδίω σε βάρο των γυναικών, ανάπτυξη. Ε, χωρίς τον προπολογισμό επίσης δεν γίνεται. Αν έχετε ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες, θα σας δώσω είτε κύριε Λάγκη εσά τι πληροφορίε, είτε στείλτε μου τα email σα. Πέτρο, σε ευχαριστώ. Πράγματι, ε, έχουμε αυτή την πρωτοβουλια ε, P20. Ε, ελπίζω να οργανωθεί του χρόνου αυτή η συνάντηση. Γιατί θα γίνει και η G20 εκεί και αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Διαφάνεια και αυτό μας χαρακτηρίζει και την Κοινοβουλευτική Ένωση και τον Κοινοβούλιο. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αν έχετε περισσότερες ιδέες για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας εν ώψη αυτής της συνάντησης P20, να μας ενημερώσετε παρακαλώ. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ και δεν τα πήγα και τόσο άσχημα από πλευράς χρόνου. Ντάνκεσεν. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σαφές ότι είναι καθήκον δημοκρατικά εκλεγμένων ε, βουλευτών να είναι πολύ ενεργοί σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι μόνο στα καθήκοντα των κυβερνήσεων, αλλά και των βουλευτών. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά, διότι ήρθατε να μας δείτε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Διατηρήστε την πίεση που ασκείτε και την ισχύ που έχετε για να αλλάξουν οι κανόνες για το κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλώς. Περνάμε τώρα στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση της ε, ad hoc αντιπροσωπείας στο Δημόσιο Φόρουμ του ΠΟΕ και στην 44η συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον ΠΟΕ στη Γενέβη 7 και 8 Οκτωβρίου του 19. Έξι μέλη πήγαν, η Καπριέλα, ο νέος αντιπρόεδρος από την Ναμίμπια, αυτό συνάντησε και είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε και τον νέο πρέσβη, Γιάο Μασάντο. Ήταν η πρώτη του μέρα που είχε μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του στη Γενέβη πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πιο καινούριο από εμά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά είχα μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Η πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ μας έκανε ένα briefing και μας μίλησε για την προετοιμασία της επόμενης υπουργικής διάσκεψης στο επίπεδο ΠΟΕ, στο πλαίσιο ΠΟΕ, που θα λάβει χώρα τον Ιούνιο του 20 στο Καζακστάν βασικό θέμα συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση κάποιων θεσμικών οργάνων και θα κάνουμε και ακρόαση στις 2 Δεκεμβρίου που θα ασχοληθούμε και θα ενημερωθούμε καλύτερα για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Μαριπιέρ Περτρέν η οποία εκπροσώπησε τη δική μας αντιπροσωπεία σε ένα πάνελ σε ένα δημόσιο φόρουμ, από πολλές πηγές έμαθα ότι τα κατάφερε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, διότι συμμετείχατε σε αυτό το δημόσιο ε, φόρουμ. Αυτά λοιπόν. Σβέν, συμπρόεδρε. Ήσουν συμπρόεδρος στην, ε, στο Steering Group. Έχεις κάτι να προσθέσεις? Ναι. Τα τρία βασικά ζητήματα που συζητήσαμε ήταν η αλληλεία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τους μηχανισμούς επίλυσης συγκρούσεων. Όλα αυτά θα τα δούμε περισσότερο και στις 11 Δεκεμβρίου. Perfect. Some other remarks from the delegation. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει να κάνει κάποιο σχόλιο? Η Marie Pierre. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Μιλήσαμε για το ρόλο των βουλευτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια και να ε, διαδώσουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνει. Ήταν ευκαιρία να διαδώσουμε το ρόλο που έχουμε στην ε, επικοινωνία μας με τον Ευρωπαίο πολίτη, γιατί μας εκλέγουν με καθολική ψηφοφορία και άρα μπορούμε να παίξουμε ρόλο παντού και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η νομοθεσία σήμερα πρέπει να ανταποκρίνεται στα μηνύματα του αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλα κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν ζητάει κάποιος άλλο το λόγο για αυτό το θέμα, Επομένω, ερχόμαστε τώρα Παρενθετικά να πω ότι η επόμενη steering committee θα λάβει χώρα, θα συνεδριάσει στις Βρυξέλλες το Μάρτιο ή το Φεβρουάριο, αν δεν απατώμε. Και μετά θα έχουμε την κοινοβουλευτική διάσκεψη πριν την υπουργική διάσκεψη στις 6 Ιουνίου στο Καζακστάν να είστε έτοιμοι και καλά προετοιμασμένοι. Περνάμε στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Αξιολόγηση του αντικτύπου που έχει η επέκταση των δασμολογικών προτιμήσεων ΕΕ Μαρόκου σε προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα. Θυμάστε, συζητήσαμε εκτεταμένα το θέμα αυτό, πώς θα ελέγχουμε τα προϊόντα τα οποία ε, προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Πώς θα εγγυόμαστε ότι τα ωφέλη της συμφωνίας θα τα δρέψουν και οι τοπικοί πληθυσμοί της Δυτικής Σαχάρας χωρίς να δεχθούμε την διεθνή κατάσταση που αφορά στην επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας. Στο ψήφισμα λοιπόν μιλούμε για ορισμένες προϋποθέσεις για τη θέσπιση μηχανισμού έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι τελωνιακές αρχές να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση για τα προϊόντα που παράγονται στη Δυτική Σαχάρα και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσθέτει το ψήφισμα ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορεί να δίδει ποιοτικά λεπτομερή στατιστικά δεδομένα και μάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές και εξαγωγές κυρίως. Θα θυμάστε ότι είναι μια συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να νοηματοδοτήσουμε αυτή την ε, συμφωνία ΕΕ Μαρόκου. Δεν περίμενα ότι τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και για να Είμαι ειλικρινή σε παρελθούσες συζητήσεις με αντίστοιχους Ευρωπαίους Επιτρόπους και με τον ίδιο. Πάντοτε εξεφράζονται αμφιβολίες για τα κατά πόσο είμαστε σοβαροί στην προσήγησή μας, κατά πόσο μπορεί αυτό να γίνει στα αλήθεια και στα σοβαρά. Σήμερα όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο μηχανισμό για αυτές τις προϋποθέσεις. Και δίνω το λόγο στον κύριο Φερνάντο Περόντε Πίκνικ από την Γενική Διεύθυνση Ταξούντ για πέντε λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Θα είμαι πολύ σύντομος για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την εφαρμογή και μετά θα απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημά σας. Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου εξ όσων γνωρίζετε. Η συμφωνία αυτή σήμερα εφαρμόζεται κανονικά. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι δεν δεχόμαστε εκθέσεις και αναφορές ούτε από τα τελωνία, ούτε από τις επιχειρήσεις, από τους εμπορευόμενους. Κανείς δεν μας λέει ότι έχει δυσκολίες να την εφαρμόσει προς το παρόν. Είμαστε σε τακτή επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά τελωνία υπ' αυτή την έννοια. Τώρα, ως προς την αξιολόγηση του αντικτύπου και ως προς την παρακολούθηση της υλοποίησης, της εφαρμογής της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Επιτρόπου Μοσκοβισή με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου, ο μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας αποτελείται από δύο συνιστώσεις. Από τη μία μεριά έχουμε την ανταλλαγή απόψεων που ε, παρέχονται με βάση τη συμφωνία και από την άλλη έχουμε βοήθεια για την παρακολούθηση των εξαγωγών. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή γίνεται βάση συμφωνίας με στόχο να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της συμφωνίας στην αηφόρο ανάπτυξη. Ε, να αξιολογήσουμε τη συμφωνία σε σχέση με το σχέδιό της για τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας αλλά και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η Επιτροπή στην πρότασή της στις 20 Σεπτεμβρίου που βρίσκεται συζήτηση με τις αντίστοιχες αρχές του Μαρόκου τα τόνισε αυτά και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας διότι οι μαροκινές αρχές θα μας δώσουν όλες τις πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε το αντίκτυπο και να καταλήξουμε σε έκθεση για τα ωφέλη που θα δρέψουμε από τη συμφωνία και με αυτή τη βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετησίως θα τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως ζητείτε ακριβώς εσείς στο ψήφισμά σας και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνεται πάντοτε το πρώτο εξάμεινο κάθε ημερολογιακού έτους. Επιπροσθέτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να αξιολογήσει επιτόπου τον αντίκτυπο της συμφωνίας και τις δραστηριότητες που διενεργούν και υιοθετούν οι εξαγωγείς και θα έχει ανταλλαγές και ε, επικοινωνίες με επιτόπου με εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και με εκπροσώπους του πληθυσμού, με πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με το μαροκινό σύστημα παρακολούθηση και εποπτεία των εισαγωγών. Πρέπει να δίδονται στατιστικά στοιχεία. Ε, και αυτό αναφέρθηκε στην ανταλλαγή επιστολών της 6ης Δεκεμβρίου, η οποία αντιγράφηκε στη συνέχεια και κοινοποιήθηκε στη δική σας Επιτροπή. Το Μαρόκο έχει θεσπίσει αυτό το σύστημα όπως έχει συμφωνηθεί και έχει δώσει πρόσβαση σε αυτό το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς δώσαμε πρόσβαση στις τελωνιακές αρχές των κρατών μελών. Και τα, οι συνιστώσεις του συστήματος είναι οι εξή. Καλύπτονται όλες οι εισαγωγές από τη Δυτική Σαχάρα με βάση την προέλευση, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία. Το σύστημα θα καλύψει όλες τις περιφέρειες του Μαρόκου διοικητικά, αλλά θα μπορούμε να ταυτοποιούμε τις εξαγωγές με προέλευση τη Δυτική Σαχάρα και όλες αυτές οι εξαγωγές εκεί θα μπαίνουν, σε αυτό το κεφάλαιο. Τα στοιχεία θα μιλούν για ποσότητα αναπροϊόν και για να αξία και τιμή αναπροϊόν με ανάλυση ανακράτους μέλος εισαγωγής. Και είναι, είναι στοιχεία που θα ενημερώνονται τακτικά κάθε μήνα σε μηνιαία βάση. Τα στοιχεία αυτά έχουν ανέβει τώρα στο διαδίκτυο, στην αντίστοιχη πλατφόρμα και είναι διαθέσιμα για το μήνα Ιούλιο, το μήνα Αύγουστο και το μήνα Σεπτέμβριο. Δική μας εκτίμηση και αξιολόγηση είναι ότι το σύστημα αυτό αντιστοιχεί με τα συμπεφωνηθέντα τον Δεκέμβριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μαροκινών Αρχών. Και όπως αναφέρθηκε στην επιστολή Μοσκοβισή, ο μηχανισμός κατά την άποψή μας πληρεί τα κριτήρια τα οποία έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο αντίστοιχο ψήφισμά του, όπου και ζητεί την παροχή αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών, στοιχείων και πληροφοριών με λεπτομέρειες που θα υποβάλλονται εγκαίρως και που θα είναι ξεχωρισμένα ως στοιχεία και ως πληροφορίες για να είναι επανάγνωστα και παρέχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά θεωρούμε. Επιπροσθέτως θεωρούμε ότι όλα αυτά συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τους μηχανισμούς που έχει η Συμφωνία για διοικητική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκών Αρχών και Μαροκινών Αρχών καλύπτεται και η δυνατότητα να, να επαληθεύσει κανείς ανα πάσα στιγμή την αληθινή προέλευση των προϊόντων που εξάγονται από τη Δυτική Σαχάρα. Άρα, κατά τη γνώμη μας, ο συνδυασμός αυτών των δύο συστημάτων, του Ευρωπαϊκού και του Μαροκινού, θα μας δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορούμε να ελέγξουμε ανα πάσα στιγμή κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Τελωνιακή Νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ποια είναι η γνώμη της εισηγήτριας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή που έδωσε όλες αυτές τις ε, προφορίες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που είπατε ήταν αρκετά ασαφή. Ε, γιατί η δική μας την ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έτσι μια εικόνα για την ιχνηλασιμότητα σε αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει μία μέθοδος συχνή λασιμότητας. Υπάρχουν απαραίτητες πληροφορίες και τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκούν αρκούν για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ποια είναι σήμερα η άποψη του σε πληθυσμού σχετικά με όλες αυτές τις πληροφορίες. Γνωρίζεται άραγε κατά πόσο να έχει προκύψει κάποιο όφελος ε, στην τοπική κοινωνία. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που δίνονται είναι σαφείς και σωστές το είπατε αυτό, αλλά θέλω να ξέρω ποια είναι ακριβώ η αξιολόγηση επιτροπή από αυτού. Και πίσω από αυτά τα στατιστικά δεδομένα, ε, η προστιθέμενη αξία που ήταν μια υπόσχεση υπάρχει, έχει προκύψει, γιατί ε, η συμφωνία έλεγε θα έπρεπε να είναι σίγουρο ότι οι χαμηλότερες τιμές θα ήταν προς όφελος του ντόπιου πληθυσμού. Έχουμε στοιχεία, έχουμε αξιολόγηση και γνωρίζουμε κατά πόσον ε, αυτή η συμφωνία στηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Και αν δούμε λιγάκι και στο μέλλον, μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι διαπραγματεύσεις ε, για ε, εμπορική και συμφωνία εμπορικών ανταλλαγών. Τα μαθήματα που μάθαμε μέχρι τώρα για το μέλλον, για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, ποια ακριβώς είναι αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρου ε, του ΕΛΚ Αντρέ Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, στις αρχές αυτού του έτους η Επιτροπή στήριξε την πρόταση να επεκταθούν οι προτιμήσεις της συμφωνίας και σε προϊόντα που παράγονται ε, στην ε, Σαχάρα προς όφελος του ντόπιου πληθυσμού. Εμείς στηρίξαμε όλα αυτά για να επανέλθουν οι προτιμησιακές δεσμολογικές συμφωνίες με τη Δυτική Σαχάρα. Το Κοινοβούλιο θέλει θέλησε να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός που θα ισχύει ε, για τα κράτη-μέλη και για τις δασμολογικές αρχές θα πρέπει όμως να δίνει τη δυνατότητα σε αυτές να έχουν πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες. Όπως προτείνεται λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το Μαρόκο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέτυχαν μια συμφωνία που αφορά στον ορισμό του μηχανισμού που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να αξιολογεί το εσωτερικό σύστημα δεδομένων του Μαρόκου για προϊόντα που εξάγονται από τη Δυτική Σαχάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρόμεθα που το Μαρόκο τήρησε την υπόσχεσή του ε, και έφτιαξε μια πλατφόρμα που προσφέρει επικαιροποιημένες πληροφορίες για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με λεπτομέρειε εταιρείες, εξαγωγές σε όγκο, ε, σε γραμμές, δασμολογικές γραμμές, αναχώρα προορισμού ε, και εξαγωγές αναπεριοχή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σχετικά με την Επιτροπή περί της ε, συνεργασίας των δύο χωρών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμφωνίας και επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή πότε περιμένετε ότι θα υπάρχει η πρώτη αξιολόγηση με βάση το μηχανισμό, με βάση το μηχανισμό που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες από τις 6 Ιουλίου του 2019. Για το Renew... Τεσέγλ με λένε, Τεσέγλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που είναι σημαντική για το Ευρωκοινοβούλιο. Να συμπληρώσω λίγο αυτό που είπαν οι δύο προλαλήσαντες εισηγητές. Αυτό το οποίο ξεκάθαρα έχει ζητήσει από την προηγούμενη θητεία το Κοινοβούλιο είναι να έχει ενημέρωση για την αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ Ένωσης Μαρόκου ποτέ δεν είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, τουλάχιστον έχουμε κάποιο ε, επίπεδο ενημέρωση πλέον για την πρόοδο. Από την ομάδα Renew ε, θα σας εκφράσω την υποστήριξή μας ε, προς τη διαδικασία αυτή. Και επίσης θέλουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με την επέκταση της συμφωνίας με τα προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα για να δούμε πώς αυτή θα επηρεάσει τα διάφορα μέρη Συνολικότερα θέλουμε να ε, πενθυμίσουμε την σημασία των σχέσεων της Ένωσης με το Μαρόκο, ένα ιστορικό εταίρο, σημαντικό ιδίως για τα γεωργικά ζητήματα. Και για να ολοκληρώσω, ένα άλλο σημαντικό θέμα για εμάς είναι το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας, που πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής λύσης υπό την πλήρη αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Δεν χρειάζεται εμείς εδώ να συζητάμε διαμακρών στην Επιτροπή μας το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Αρκεί να είμαστε βέβαιοι ότι οι επιλογές μας θα ωφελήσουν όλες τις πλευρές. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους πράσινους, η κυρία Μπρικμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, κάποιες ερωτήσεις αφού σα ευχαριστήσω που βάλετε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, είναι σημαντικό για του πρασίνου και η συνάδελφο αλλά έχει συνεργαστεί. Μάλλον έχει εργαστεί πολύ για αυτό το θέμα. Κάποιε ερωτήσει. Κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο υπάρχει υποχρέωση αναφοράς ξεκάθαρα ε, της καταγωγής του προϊόντος. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει αυτή η μνήμα για τα πρώτα από τη Δυτική Σαχάρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αξιολογεί τις τρέχουσες πρακτικές. Δεύτερη ερώτηση. Γεωγραφικά όρια στις νότιες επαρχίες που δεν είναι το ίδιο γιατί περιλαμβάνουν μαροκινά εδάφη, δηλαδή όχι μόνο τη Σαχάρη, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν καλύπτεται και υπάρχει και ένα κομμάτι που είναι υπό τον έλεγχο του ε, Μαρόκου. Τι προβλέπεται να γίνει. Και τέλος, τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα, αλλά από εδάφη εκτός ελέγχου του Μαρόκου, αυτά δεν ωφελούνται από τις ε, προτιμησιακές τιμές, προνομιακές τιμές. Τι θα γίνει λοιπόν, μιλάμε για διαφορετική μεταχείριση στο έδαφος του ίδιου κράτους. Επίσης, αρμόδια αρχή για την έκδοση επιστοποιητικών εισαγωγή αυτών των Πέντε στην Ευρώπη, ποια είναι. Ευχαριστώ. Και εμείς ε, και τώρα ε, εκ μέρους της ε, ο πρώην συγκητής μας για το Μαρόκο, κύριο Μορέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Άρα μιλάω επί προσωπικού, μιλάω εξ ονόματός μου μόνο για να το ξεκαθαρίσω αυτό, χωρίς να, να θέλω να πω ότι δεν υπάρχει συνεργασία μαζί μας. Εντίθετα υπάρχει και συνεννόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Είναι μια από τις λίγες σταθερές ε, χώρες περιοχής στο Μαρόκο και η εταιρική σχέση που έχουμε με αυτή τη χώρα είναι στρατηγική σημασίας. Όπως είπα ε, ο συνάδελφος από το Ρινιού, το θέμα εδώ δεν είναι ε, να συζητάμε το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Παρότι νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΓΑΜΑ των Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσει τα ε, μέρη να καταλήξουν μια βιώσιμη λύση κτλ. κτλ. Τα επιχείρηματα τα ξέρετε. Πολύ εργαστήκαμε στη τελευταία θητεία μαζί με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Σε συνέχεια και των προϋποθέσεων ε, που έθεσε το δικαστήριο θέλουμε να υπάρξει όφελος για τους πληθυσμούς. Ένα αυτό. Αλλά μου φαίνεται αόριστο ακόμη. Δεν καταλαβαίνω απόλυτα ο μηχανισμός αυτός πώς θα οδηγήσει σε αυτό. Δεύτερον, συγκεκριμένα θέλουμε να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών με τις τελωνικές αρχές του Μαρόκου. Η Κομισιόν θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένη γι' αυτό. Πώς, πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Και τρίτον, η απόφαση της Επιτροπής Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου για την αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτής της συμφωνίας σε ποιο βαθμό βρίσκεται και αυτό που και η Καθλήν Φον Μπρέμπτ νομίζω. Μεθοδολογία, ηχνηλασιμότητα. Πολλής λόγος έχει γίνει και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω. Δεν έχω καταλάβει όμως ακριβώς. Επειδή ξεκινάμε τώρα ε, τη νέα θητεία, καλό είναι να ξεκινήσουμε από τη σωστή βάση και θα ήθελα η Κομισιόν να μας δώσει κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Και πριν ε, λοιπόν ε, δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας να λάβει το λόγο, ο κύριος Κοτσολίνο, για δύο λεπτά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, φαντάζομαι ε, ότι ισχύουν όλα αυτά τα οποία είπαν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά ε, στο Μαρόκο αυτή η περιοχή είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, στο Μαγκρέπ, και έχουμε μια πολύ καλή σχέση ε, όσον αφορά ε, τις κοινοβουλευτικές μας επαφές. Τις επόμενες εβδομάδες ε, θα προχωρήσει ο κοινοβουλευτικός διάλογος και αυτό κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια σημαντική συμφωνία για τους κατοίκους του Μαρόκου και για την Ευρώπη. Είναι μια συμφωνία σημαντική λόγω των σχέσεων που έχουμε το Κοινοβούλιο του Μαρόκου και λόγω των εμπορικών ανταλλαγών. Πρέπει λοιπόν να επιβεβαιώσουμε τη θέληση και βούληση για συνεργασία και μετά βέβαια να δούμε ε, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ε, καθώς ε, προχωράει η συμφωνία. Ενδεχομένως να διορθώσουμε και τα στοιχεία, να γνωρίζουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καθόρισε το πλαίσιο, σημαντικό αυτό, αλλά θα πρέπει πάνω απ' όλα να καθορίσουμε αντικειμενικά κριτήρια για τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στον, στους κατοίκους ε, του Μαρόκου και της Δυτικής Σαχάρας. Σας είπα όμως ότι εδώ δεν πρέπει να υπάρξει ε, μια εξέλιξη όπου θα ωφεληθούν άλλοι. Δεν είναι εδώ ο κατάλληλος χώρος να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ε, πρέπει να έχουμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα ωφελήσει αυτή η εμπορική συμφωνία τον τόπιο πληθυσμό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι να ε, έχω περισσότερες λεπτομέρειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κατανοήσω με βάση τις εμπειρίες μας τι θα γίνει στο μέλλον. Ε, τι μπορεί να υπάρξει ε, τι ε, νέες συμφωνίες μπορούμε να συνάψουμε, καινοτομίε σε αυτή τη διαδικασία, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά όλα πρέπει να τα προσπαθήσουμε γιατί βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη ε, κατά την προηγούμενη θητεία παίξαμε ε, πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, μαγάρι να είχαμε εμπορικέ συμφωνίες με όλη τη Βόρεια Αφρική, τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες όπως αυτές που έχουμε με το Μαρόκο. Θέλω λοιπόν να καλέσω την Επιτροπή να μας πει τι είδους νέα μέτρα πρέπει να λάβουμε και για να εφαρμοστεί αυτή η εμπορική συμφωνία και για να γίνει και η κατάλληλη αξιολόγηση. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε και μια κοινή συνεδρίαση με την κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία με τις χώρες Μαγκρέπ, κυρίως με το Μαρόκο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που ε, μας είπατε σήμερα και τα παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, Πενιέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω την αξία που έχει η συμφωνία με το Μαρόκο και η δέσμευση που έχουν αναλάβει και τα δύο μέρη, και η Επιτροπή και οι Μαροκινές Αρχές, για να εκπληρώσουν το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θυμάμαι, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξουμε σε μηχανισμό που να μπορούσε να κάνει αξιολόγηση της συμφωνίας και ότι πράγματι τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας θα μπορούσαν να δρέψουν τις δασμολογικές προτιμήσεις που δίδονται ε, στο Μαρόκο. Όπως και οι μαροκινές αρχές άλλωστε. Και μας εξηγούσαν τότε ότι υπήρχαν διάφορες δυσκολίες για να συγκεντρωθούν πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται ξεπεράστηκαν αυτές οι δυσκολίε αυτές. Θέλω να ρωτήσω γιατί ήταν τόσο ανυπέρβλητες στην προηγούμενη θητεία και πώς καταφέρατε να τις ξεπεράσετε και πώς συγκεντρώνετε τώρα τα στοιχεία. Θέλω επίσης να τονίσω το εξή. Παρόλο που στην απόφαση του Συμβουλίου έχουμε στοιχεία σε αιτήσια βάση οι μαροκινές αρχέ θα μα τα στέλνουν σε μηνιαία βάση και αυτό είναι πολύ θετικό βήμα. Έχω το εξή συγκεκριμένο ερώτημα να απευθύνω στην Επιτροπή. Στην πρόταση απόφαση του Συμβουλίου γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση του ενδυνάμει αντικτύπου της Συμφωνία στις εμπορικές ροέ τη παρελθούσε. Στις προβλέψεις όμως που κάνετε για τις μελλοντικές εμπορικές ροές, για την αλία, για τα φωσφορικά προϊόντα, και άλλα και τα γεωργικά. Πώς ακριβώς το κάνετε, δηλαδή οι προβλέψεις που έχετε για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο αντιστοιχούν με την αξιολόγηση αντικτύπου και τις, ε, τα στοιχεία που είχατε προβλέψει, τα στοιχεία του τελευταίου τριμήνου. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ θετικό ότι διευκολύνουμε τώρα και έχουμε ένα σύστημα πληροφόρησης όμως πρέπει να μπορούμε να το ελέγχουμε, να δούμε αν είναι αρκετό. Και αν τα αποτελέσματα του συστήματος αυτού πράγματι θα μας κάνουν να εγγυόμαστε ότι θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτή τη συμφωνία οι κάτοικοι της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, όπως και οι συνάδελφοι προηγουμένως και εγώ είμαι ευχαριστημένη κυρίως ε, διότι ε, το Μαρόκο ανταποκρίθηκε ταχύτατα στις ανησυχίες μας σχετικά με την γεωγραφική χνηλασιμότητα των προϊόντων που εξάγονται στην Ευρώπη. Ε, μπορούμε λοιπόν να εντοπίσουμε την προέλευση των προϊόντων ε, και το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά ε, για τους Μαροκινούς για τη Δυτική Σαχάρα ο μηχανισμός ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικό. Σήμερα εκφράζονται κάποιες απόψεις επ' αυτού, αλλά θεωρώ ότι η Επιτροπή ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορούμε και να τοποθετηθούμε, θα διαθέσει τα απαραίτητα στοιχεία. Εύχομαι λοιπόν να μην φτάσουμε σε πολιτική χειραγώγηση ε, της απόφασης ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και γενικότερα του μηχανισμού, γιατί όλοι εύχονται να υπάρχει μία άποψη που να τους εκφράζει όλους στη Δυτική Σαχάρα. Απ' την άλλη όμως σας λέω ότι το εμπορικό θέμα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχωρίζεται από τις γενικότερες εξελίξεις. Ο κύριος Κάνας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε τη διεύρυνση, τον αντίκτυπο της διεύρυνσης των δασμολογικών προτιμήσεων για να συμπεριληφθεί και η Δυτική Σαχάρα. Καλό θα είναι να ξέρουμε πώς επηρέασε και τα τοπικά προϊόντα. Εν πάση περιπτώσει, κάπως να ασχοληθεί η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή με τους Ευρωπαίους παραγωγούς, έτσι δεν είναι. Στην Αλμερία, στην Ισπανία, είμαστε η μεγαλύτερη παραγωγή ντομάτας. Και εγώ τους ρώτησα εκεί αυτή η κατάσταση, τι αντίκτυπο είχε σε εσά, αλλά ε, άκουσα από αυτά που έρθει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει. Όταν ακούω τους παραγωγούς δεν μας λένε την ίδια αφήγηση, μας λένε κάτι πολύ διαφορετικό, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι υπάρχει λαθρεμπορία μαροκινών ντοματών μαροκινή ντομάτα που πλημμυρίζει την ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχει χαλαρότητα στου ελέγχου. Μιλούμε για χιλιάδε τόνου που μπαίνουν ως ευρωπαϊκή ντομάτα και υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκή ντομάτα, αλλά είναι από το Μαρόκο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο ε, εισάγονται παράνομα ντομάτες από το Μαρόκο και θα μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά πόσο εισάγονται παράνομα ε, ντομάτες από τη Δυτική Σαχαρά. Είμαστε σοβαροί να σκεφτούμε και τους Ευρωπαίους παραγωγούς, οι οποίοι μας λένε ότι η αγορά τους από οροκυπευτικά πλημμυρίζεται από ε, παραγωγούς που κάνουν λαθρεμπόριο, που βαφτίζουν μαροκινές ντομάτες για ισπανικές ή ευρωπαϊκές και θα πρέπει οι συμφωνίες να τηρούνται. Όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι πολύ απλά. Να μην διαβάζουμε μόνο τα στατιστικά στοιχεία των μαροκινών αργών, να διαμιλήσετε και με τους ε, ντόπιου παραγωγούς που αποτελούν και την ευρωπαϊκή βιομηχανία άλλωστε. Τώρα, αν μέλημά μας είναι να ωφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός, επενεταίο βέβαια, ε, τότε δεν βλέπω γιατί στις εκθέσεις ε, να στηρίζεται περισσότερο ο μαροκινός πληθυσμός. Επομένως, θεωρώ το εξής. Επαναλαμβάνω, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ιχνηλασιμότητα της μαροκινής ντομάτας, θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ιχνηλασιμότητα της ε, ντομάτας της Δυτικής Σαχαράς. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει επιθεωρητές για να δει κατά πόσο και ελεγκτές στηρούνται όχι μόνο τα δασμολογικά και τα τελωνιακά και τα εμπορικά, αλλά και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κατοχή αυτών των εδαφών. Και θα το κάνουν οι μαροκινές αρχές και θα τις πιστεύουμε. Το εμπόριο δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο. Πρέπει να εγγυαόμαστε τους στόχους αλλά και την ισότιμη μεταχείριση των Ευρωπαίων παραγωγών. Εγγυόμαστε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και εγγυόμαστε και τις νέες ε, συνθήκες και διατάξεις για τη φυτογενομική προστασία και να εγγυηθούμε ότι θα ανταγωνίζονται όλοι υπό τις ίδιες συνθήκες. Να μην αξιοποιεί το βασίλειο του Μαρόκου μια ανθρωπιστική κατάσταση για ε, λόγο εμπορικό και για να εκμεταλλεύεται και να δρέπει οικονομικό όφελος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χαουτάλα, παρακαλώ. Um, I find it... Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κατανοώ όλο αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι υποκριτικό το να λέμε ότι πρέπει να μιλάμε μόνο για την εμπορική πολιτική και άλλοι να ασχοληθούν με την εξωτερική πολιτική. Ε, η εμπορική πολιτική πρέπει να ε, δράζεται σε μια νομική βάση και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι το Μαρόκο δεν μπορεί να έχει κυριαρχία επί της Δυτικής Σαχάρας. Και ρωτώ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια είναι η νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι εισαγωγεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέχονται τις εισαγωγές προϊόντων από τη Δυτική Σαχάρα. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ενημερωθούμε για το πώς η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ραμπάτ, πώς αυτή η αντιπροσωπεία χειρίζεται τη συμφωνία και την εφαρμογή της, ε, πώς το κάνει αυτό με τις αρμόδιες αρχές του Μαρόκου. Ε, γιατί αν κάνουμε μία σύγκριση. Ας δούμε, οι Ευρωπαίοι στη, εκπρόσωποι στη Ρωσία και το Ισραήλ, αυτοί δεν μπορούν να αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα στην ε, Κρυμαία και στην Δυτική Όχθη. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν εσείς ε, πώς ακριβώς θέλετε να προχωρήσετε σε αυτό το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Η δική μου ομάδα είχε κάποιες επιφυλάξεις και γι' αυτό καταψηφίσαμε και οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν. Γιατί ήδη αυτή την εβδομάδα ακούσαμε ότι υπάρχουν ε, σοβαρές ε, διώξει ακτιβιστών ανθρωπίνων δικημάτων στη Δυτική Σαχάρα οι οποίοι επέκριναν τι αρχές του Μαρόκου. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε τόσο αφελείς όσον αφορά το μηχανισμό ο οποίο φαίνεται να έχει εγκατασταθεί και δεν ακούσαμε καθόλου το ποιε είναι οι επιπτώσει αυτού του μηχανισμού. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ την Επιτροπή και παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε τελευταίος ε, ερωτών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 ο κύριος ε, Σουστέρ Και εγώ πρέπει να σας πω ότι με λιγάκι που μας λέτε συνέχεια ότι ε, θα εγκατασταθεί ένας ε, μηχανισμός στις αρχές του έτους όταν όλο αυτό ήταν πίδικο έμοιαζε ότι τον Μάρτιο-Απρίλη θα εγκριθεί ο μηχανισμός και σήμερα υποτίθεται θα είχαμε και την πρώτη έκθεση για το θέμα ήταν φλέγον και ρωτώ εγώ κατηγορηματικά παρακαλώ επιτέλους πότε θα μας δώσετε αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την προέλευση των εισαγωγών μας από το Μαρόκο. Ε, ποια είναι η περιφερειακή τους προέλευση, ε, τι ποσοστό καταλαμβάνουν στο σύνολο των εξαγωγών και ε, ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας επωφελείται και αν ναι, σε ποιο βαθμό. Αυτό θέλαμε να μάθουμε. Ε, υπήρξε η αδιαμφισβήτητη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τότε τα πράγματα μας τα είχατε παρουσιάσει λιγάκι διαφορετικά και γι' αυτό έχω θυμώσει λιγάκι. Ε, Επίση, ε, να σας πω ότι θεωρώ ότι πρέπει εδώ να έχουμε τους σωστούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί όλη αυτή η διαδικασία της ε, διαμεσολάβησης αναχαιτίστηκε γιατί ε, παραιτήθηκε ο κύριος Κέλλερ το Μάιο. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία επίλυσης της διένεξης. Ίσως λοιπόν ε, να έχουμε εδώ κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να είναι σε θέση να μας ενημερώσει. Αν δεν είναι κανείς που να είναι σε θέση να ενημερώσει, παρακαλώ να μας ενημερώσετε εκ των υστέρων σε γραπτή μορφή. Περόντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο θέματα. Το ένα είναι η χνηλασιμότητα και το άλλο είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Σχετίζονται τα θέματα αυτά, αλλά και ενδιαφέρον. Όσον αφορά την χνηλασιμότητα, όσο συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ιδέα είναι να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι απόλυτα συμβατά και συμμορφωμένα με την ε, δική μας την νομοθεσία. Υπάρχουν στοιχεία για τις εισαγωγές και σε περίπτωση αμφιβολίας μπορεί κανείς να ε, επαληθεύσει, να εξακριβώσει την προέλευση των προϊόντων. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύστημα πληροφοριών που δίδονται από το Μαρόκο σε συνδυασμό με τον μηχανισμό δεσμολογικής συνεργασίας που έχει ε, εγκατασταθεί με βάση τη συμφωνία. Βέβαια, αυτό είναι διαφορετικό. Είναι βέβαια συμπληρωματικό στην αξιολόγηση των επιπτώσεων, για την οποία αξιολόγηση το βασικό εργαλείο δεν είναι τα στατιστικά δεδομένα, είναι και αυτά, αλλά βασικός και καθοριστικός είναι ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών, όπως προβλέπει η συμφωνία. Με βάση αυτό το μηχανισμό το Μαρόκο υποχρεούται να καταθέτει όλα τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, την χρήση των φυσικών πόρων, οτιδήποτε χρειάζεται για να αξιολογήσει κανείς τις επιπτώσεις. Και βεβαίως για να αξιολογηθούν επιπτώσεις είναι σημαντικό να υπάρχουν και στατιστικά δεδομένα για τις εμπορικές ανταλλαγές. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Τα δεδομένα που δίδονται από το Μαρόκο είναι ικανοποιητικά μέχρι Τώρα ε, πρέπει να σας πω ότι είναι λεπτομερή, ότι αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία έχει δεχτεί το Μαρόκο και ε, σε αυτά που ζήτησε το Κοινοβούλιο μέσα από το ψήφισμά του. Δεν κάναμε βέβαια επαλήθευση των ε, στοιχείων, αλλά με τις πληροφορίες μέχρι τώρα φαίνεται ότι πράγματι τα στοιχεία βαδίζουν προς την ε, κατεύθυνση που είχαμε καθορίσει εμείς ε, σχετικά με, το, με τις εξαγωγές ε, από τη Δυτική Σαχάρα. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έχουμε μια τελική αξιολόγηση γιατί τα στοιχεία είναι πολύ φρέσκα. Μόλις πριν από τρεις μήνες ε, συνήφθη η συμφωνία και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς αν είχαν θετικές επιπτώσεις στον τόπιο πληθυσμό. Για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Να πω επίσης ότι για την Επιτροπή ε, Νομίζω ότι είναι δυνατόν να προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία. Βεβαίως, ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει αμέσως, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που ανταλλάσσουμε πληροφορίες το 2019 δηλαδή. Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών θα ε, συνεχιστεί το 2020 και τα διαρκέσει πάρα πολλούς μήνες. Και μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μόνο τότε θα μπορούμε να σας δώσουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Ε, βεβαίως, αν το ζητήσετε, μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες ε, που παίρνουμε από την Τράπεζα Δεδομένων του Μαρόκου, ε, να έχετε κι εσείς, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα στα ερωτήματα που αναφέρονται στην προέλευση των προϊόντων. Η συμφωνία δεν λέει τίποτα όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων. Η συμφωνία ε, αναφέρεται στο ότι είναι απαραίτητο ε, τα προϊόντα να σέβονται τους κανόνες της προέλευσης. Τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα ε, να ε, σέβονται τις προδιαγραφές για να επωφελούνται και από τις δασμολογικές ε, προτιμήσεις. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο θέμα δασμολογικό, είναι θέμα που έχει σχέση περισσότερο με την εσωτερική αγορά. Ετέθη κατόπιν ένα ερώτημα σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις επαρχίες του Μαρόκου και τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω επ' αυτού είναι ότι όλες τις πληροφορίες που δίδονται από το Μαρόκο ε, για τις επαρχίες όλα αυτά ε, ταυτίζονται πλήρως με τα προϊόντα που εξάγονται από τη Δυτική Σαχάρα. Παράδειγμα, ε, επαρχία Γκέρμιγκ βρίσκεται κατ' ουσίαν στο Μαρόκο. Έχει όμως και ένα μικρό κομμάτι στη Δυτική Σαχάρα. Και από εκεί ε, από το κομμάτι της Δυτικής Σαχάρας δεν υπάρχουν εξαγωγές γιατί αυτό είναι ε, μέσα στην έρημο, δεν έχει από εκεί εξαγωγές. Αυτό ήταν έτσι ένα μικρό παράδειγμα που ήθελα να σας αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά τις ε, περιοχές που είναι εκτός ελέγχου των μαροκινών αρχών. Ε, δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν αρχές. Δεν υπάρχουν αρχές που να μπορούν να πιστοποιήσουν ε, προέλευση προϊόντων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να το πούμε κιόλα ότι σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν προϊόντα που να μπορούν να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όσον αφορά τις ε, ανησυχίες του κ. Κάνια ε, σχετικά με την έλλειψη των ελέγχων, ε, δεν έχουμε πληροφορίες για το να υπάρχουν εισαγωγές που να βασίζονται σε απάτη ε, από το Μαρόκο. Δεν υπάρχουν ε, εισαγωγές ε, που να έχουν παρακάμψει κάτω κάποιες φυτογειονομικές διατάξεις, αλλά αν έχετε κάποιες πληροφορίες, πολύ ευχαρίστω να το ελέγξουμε το θέμα και αυτό μπορούν να το πράξουν οι συνάδελφοί μας που είναι αρμόδιοι για τις αγορές, η Γενική Διεύθυνση Άγκρη, από με τη Γενική Διεύθυνση Τάξουντ. Όσον αφορά τώρα στις επιπτώσεις επιτόπου, εμείς δεν θα κάνουμε επιθεωρήσεις, ελέγχου σε ξένα εδάφη, δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Επιτροπή, αλλά οι αρχές του Μαρόκου ε, είπαν ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτες να επισκεφθούν τη Δυτική Σαχάρα και να έχουν επιτόπου αν συζητήσεις με τους ντόπιου παραγωγούς. Άρα δηλαδή αν θέλετε θα υπάρξει ε, κάποια συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόπου θα γίνουν όλα αυτά. Όσον αφορά τώρα τη νομική βάση για την αναγνώριση ε, των ε, πιστοποιητικών, η νομική βάση είναι κατ' ουσίαν η ίδια συμφωνία. Συνήψαμε μία συμφωνία με το Μαρόκο, γιατί αυτή είναι η μόνη αρχή που μπορεί να πιστοποιήσει και να σεβαστεί τους κανόνες της προέλευσης. Αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου, ε, τώρα πλέον εναπόκειται στο δικαστήριο μετά από το αίτημα του, τον Πολυσάριο κατά της συμφωνίας να προχωρήσει το δικαστήριο. Ε, το θέμα αυτό νομίζω θα συνεχιστεί και θα ενημερωθούμε. Ε, τώρα, αυτό που ενδιαφέρει τις δασμολογικές αρχές είναι ε, το κατά πόσον αυτά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Μαρόκο, κατά πόσον είναι αυθεντικά και κατά πόσον καλύπτουν τις προδιαγραφές μας. Όλες οι πληροφορίες που έχουμε τίνουν προς την κατεύθυνση ότι πράγματι έτσι είναι. Και τέλος, όσον αφορά στο πότε θα έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για τις εξαγωγές από τη Δυτική Σαχάρα. Όπως σας είπα, το ερώτημα τέτοιο από τον κύριο Σούστα, οι πληροφορίες αυτές μας δίδονται σε ε, τακτική βάση ε, και γι' αυτό και εμείς αν το θέλετε να σας τη δίνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να σας καταθέσουμε λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων, γιατί όπως σας είπαμε δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ε, επίστηνα ιδιαίτερα, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ούτε κι εγώ επίστην. Δεν θέλω να είμαι γιατί ξεκινάει η νέα θητεία και θέλουμε καλές σχέσεις. Είναι ένας φάκελος πολύ σημαντικός με ένα στρατηγικό εταίρο. Και καλά έκανε και μπήκε το θέμα στη μέση διάταξη. Ακούγοντα όμω τι λέει η Κομισιόν, δεν ξέρω, ίσω είναι πολύ νωρί να μα δώσει πραγματικά στοιχεία η Κομισιόν ε, για το τι συμβαίνει επί τόπου. Μέχρι τώρα Πίστευα ότι καλό θα ήταν να έχουμε πολύ σύντομα τη συγκρότηση της πρώτης ομάδας παρακολούθησης για να έχουμε εντελεχείς και βαθ... διεξοδικές συζητήσεις για την ειχνηλασιμότητα, τα δεδομένα, τα στατιστικά, τη μελέτη αντικτύπου, αλλά και το θέμα που σας έθεσα και δεν απαντήσατε, ίσως γιατί δεν έχετε απάντηση, δηλαδή ποιο είναι ακριβώ ο αντίκτυπο στη Δυτική Σαχάρα και ποια είναι η προστιθέμενη αξία στη Δυτική Σαχάρα, που ήταν ένα μείζον ε, ε, κομμάτι του ψηφίσματος προηγούμενου κοινοβουλίου. Και δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι θα καταθέσετε αναλυτική έκθεση στο πρώτο εξάμεινο του 2020. Έτσι για να ε, σιγουρευτώ. Είπατε ότι θα δημοσιοποιήσετε την πρώτη πραγματική έκθεση για το θέμα στο πρώτο εξάμεινο του 2020 Απάντηση. Μπορεί να απαντήσει, μάλλον είναι πρόεδρος, μπορείτε να απαντήσετε. Να, ακου, να απαντήσω όλα τα ερώτημα, τα μαζί. Πρώτον, να πω ότι θα γίνει η έκθεση, αλλά αφού συλλέξουμε πρώτα όλες τις πληροφορίες από τις αρχές του Μαρόκου, που θα πρέπει να τις έχουμε στο πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά θα έχουμε επισκέψει επιτόπου, αξιολόγηση και μελέτη αντικτύπου. Η μελέτη αντικτύπου δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, επιτευχθεί μέσα σε μια εβδομάδα ή μέσα σε ένα μήνα. Σε ό,τι διαφορά αφορά το ερώτημα για τι προσδοκίες σας να έχετε τώρα τη μελέτη αντικτύπου, σας υπενθυμίζω πολύ απλά τι λέει το ψήφισμα. Ζητεί ετήσια αξιολόγηση από πλευράς κομισιών θα είναι ετήσιες αυτέ οι αξιολογήσεις αφόσον έχουμε στη διάθεσή μας επαρκεί πληροφορίες που θα τι έχουμε αξιολογήσει. Πριν όχι. Βγαίνω από τα παπούτσια μου, για να μην πω βγαίνω από τα ρούχα μου, ε, από αυτά που λέτε. Ε, γιατί εδώ στο Κοινοβούλιο που το συζητήσαμε και συμφωνήσαμε, ε, δείξαμε εμπιστοσύνη απέναντι στην Κομισιόν. Είχαμε πολλές συζητήσεις με τον κύριο Μοσκοβισή και τον εμπιστευτήκαμε. Πιστέψαμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε έναν ακριβή μεχανισμό με αξιόπιστα στοιχεία. Και έρχεστε εσείς εδώ τώρα και λέτε, ε, και τι έγινε τώρα να είναι ένα χρόνο αργότερα. Κάτι θα έχουμε, ε, κανείς δεν ξέρει πότε, κανείς δεν ξέρει πώς. Ε, πραγματικά αυτό είναι λίγο απογοητευτικό. Αν ήξερα θα μας δίνετε αυτή την απάντηση ένα χρόνο πριν, δεν θα το είχα δεχτεί αυτή τη συμφωνία με την Επιτροπή για να μην ειλικρινείς. Εμείς θέλουμε έναν σαφή μηχανισμό, σύντομα, με αξιόπιστα δεδομένα. Αλλιώς Είμαι βέβαιος ότι θα αναλάβει δράση το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, καλός ή μάλλον κακός, αλλά τέλος πάντων. Έτσι ολοκληρώνεται το σημείο αυτό για σήμερα, αλλά φυσικά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα στην ε, αρμόδια ομάδα παρακολούθηση και θα το ξανασυστήσουμε και στην Επιτροπή μας σύντομα. Πηγαίνουμε στα σημεία 17 και 18 της ημερησιάς διάταξης. Κοινή συζήτηση για το βόλιο κρέας υψηλής ποιότητας προερχόμενο από τη ΣΥΠΑ. Ένα θέμα που το συζητήσαμε ήδη όταν συνεδριάσαμε στις 2 Οκτωβρίου. Και τώρα αλλάζω ιδιότητα και από πρόεδρος γίνομαι εισηγητής. θα υπάρξει έγκριση, ε, σύμφωνη γνώμη δηλαδή για τη διαδικασία αυτή. Ε, θα ακολουθηθεί μια κάπως έκτακτη διαδικασία. Γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε συνοδευτικό ψήφισμα. Regarding Σε ό,τι αφορά ε, την απόσταση που μας χωρίζει από τη ΣΥΠΑ, και επειδή είμαστε στην εποχή των παγετώνων αυτή τη στιγμή με την ε, χώρα αυτή, θελήσαμε να προσπαθήσουμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση, γνωρίζοντας βέβαια ε, ότι το βόλιο κρέας υψηλής ποιότητας δεν έχει άμεση σχέση με τις επιδοτήσεις ε, στις αεροπορικές μεταφορές ή στις ελιές από την Ισπανία ή στο χάλιβα και το αλουμίνιο τουλάχιστον όχι άμεσα. Όμως, παρόλα αυτά, υπάρχει η σχετική ε, διαμάχη σε επίπεδο ΠΟΕ σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εισαγωγή σε βιώιο κράτος με ορμόνες χάσαμε και αποφασίσαμε στις ε, χώρες ε, να δώσουμε αθασμολόγητη προσφορά. 45.000 τόνους ε, υψηλής ποιότητας βόηου κρέατος. Το αμερικανικό βόηο κρέας κατά το παρελθόν περιλαμβανόταν στην ποσόστοση, αλλά το μερίδιό του ήταν υποτιμημένο. Τώρα προτείναμε ένα ξεκάθαρο ποσοστό, 35.000 συγκεκριμένα είναι οι τόνοι, για τη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας υψηλής ποιότητας. Το ψήφισμά μου λοιπόν, ξεκαθαρίζω, πως αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς ε, την ε, αποκλιμάκωση των σχέσεων. Και βέβαια προσδοκάμε και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δραστηριοποιηθεί στην ίδια κατεύθυνση για να υπάρξει αποκλιμάκωση και λιώσιμο των πάγων. να δεχθούμε λοιπόν αυτές τις ε, ποσότητες κρέατος. Γιατί είπα, υπάρχουν και άλλες χώρες, η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη, που αφορώνται από τον ίδιο κανονισμό και δέχονται την αλλαγή ποσόστοσης. Και έρχομαι στην Κομισιόν, την καλώ να σχολιάσει την πρόταση, της προτάσεις μου, ο κύριος Χιμένεθ από την αρμόδια μονάδα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη για τις χώρες Λατινικής Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Παρεμβαίνω εδώ εκ μέρους του κύριου Κλάρκ, του διευθυντού μου, που δεν είναι όμως σήμερα στις Βρυξέλλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί διευκολύνατε το έργο μου, Πρόεδρε. Τα είπατε όλα εσείς από μόνο σας. Ό,τι έπρεπε να υποθεί ήδη λέγεται στο ψήφισμα και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι δύο-τρει διευκρινήσει και δύο-τρία πράγματα έτσι πιο δεξοδικά να σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα ότι ναι, ελπίζουμε να ε, είναι αυτό το τέλος ε, μιας διαμάχης που κρατεί καιρό τώρα. και πάντα εντός των ορίων της διαπραγματευτικής εντολής που δόθηκε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ιδίω θέλω να τονίσω το γεγονός ότι ακριβώ με αποτέλεσμα, μάλλον αυτής της, ε, ως αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής δεν θα έχουμε αυξημένη ποσόστοση, για το βεβαίως παραμένει ως έχει και το μόνο που γίνεται είναι μια ανακατανομή διαφορετική, δηλαδή υποδιέρεση ε, μεταξύ των χωρών. Δηλαδή δεν αυξάνεται η ποσόστοση συνολική. Και βέβαια τα πρότυπα ποιότητα παραμένουν τα ίδια. Που σημαίνει το βέβαιο κρέας που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει υποστεί ε, επεξεργασία με ορμόνες άλλα προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω ότι για να προχωρήσουμε ε, πρέπει να εγκριθεί το σταμότερο δυνατόν ε, αυτή η ποσόστοση. Σας, σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας προς αυτή την κατεύθυνση και τέλος θέλω να υπογραμμίσω πως αυτή η προσαρμογή είναι εφικτή ακριβώς ε, χάρη στην σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων χωρών και δεν προβλέπεται αποζημίωση αντιστάθμιση στι χώρες αυτές. Ε, και θέλω να το πω για να το καταλάβουν όλοι. Δεν προβλέπεται πρόσθετη ποσότητα ή κάποια άλλη αντιστάθμιση αποζημίωση. Η, σημα... η ποσότητα παραμένει ίδια. Η ποσόστοση δεν αλλάζει. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Το ε, σχέδιο ψηφίσματός σας κύριε Πρόεδρε τα εξηγεί καλύτερα και από ό,τι θα τα έλεγα εγώ τα πράγματα. Σας ευχαριστώ γιατί διαχειριστήκατε τάχιστα το θέμα. Ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρος, φυσικά είμαστε αξιόπιστοι και πάντοτε είμαστε και ευέλικτοι στο Κοινοβούλιο για να λύνουμε προβλήματα. Σκιώδες εισηγητές. Ο Κριστόφ Χάνσεν από το ΕΛΚ. Δεν θα τα πω ισπανικά τώρα, ούτε πολωνικά, θα τα πω αγγλικά. Αντικαθιστώ τη συνάδελφό μου την Τανούτα Χούμπνερ, η οποία πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες για τη συμφωνία, καθότι ήδη είχαμε ανταλλαγή απόψεων στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ως σκιώδης εισηγητρία πάντως θέλει να τονίσει ότι είναι σημαντική η συμφωνία στο πλαίσιο των προσπαθειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει εμπορικέ εντάσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε προ τη ΗΠΑ ότι η συμφωνία αυτή θα επικυρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Επομένω, άποψη του ΕΛΚ είναι ότι θα πρέπει ε, να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να μην καθυστερήσουμε την επεξεργασία αυτού του φακέλου. Αν έχουμε συμφωνία πριν το τέλος του χρόνου, θα δώσουμε ένα θετικό μήνυμα προς τους ομολόγους μας από τη ΣΥΠΑ, ότι είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε ώστε το, τη δήλωση Γιούνκερ Τραμπ του Ιουλίου να την ε, εφαρμόσουμε στην πράξη πλέον. Ελπίζουμε να υπάρξει αίσιο πέρας, να υπάρξει σύναψη συμφωνίας ώστε αυτή η δήλωση του Ιουλίου, Γιούνκερ τράμπ του Ιουλίου του 2008 να γίνει πραγματικότητα. Και έτσι να δοθεί έτσι μια πιο θετική νότα και απόχρωση της σχέσης των δύο πλευρών. Πριν τον Ιανουάριο λοιπόν του 2020 ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει και ελπίζω στα τέλη Νοεμβρίου να ψηφίσει ολομέλεια. Είναι καλό το σχέδιο έκθεσης, άρα το ΕΛΚ δεν θέλει να γίνει κάποια τροποποίηση. Επίση, ζητούμε από τι άλλε πολιτικέ ομάδε να μην προβούν σε δραστικές αλλαγές του κειμένου, ώστε εγκαίρω και επιτυχώ να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτού του ζητήματο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σράινεμαγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. καταρχά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο με την ιδιότητά του του εισηγητή για τη σύνταξη ενό πολύ ισορροπημένου ψηφίσματος εν, μέσω εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι η συμφωνία που καταφέραμε και πετύχαμε με τις ΗΠΑ πριν το καλοκαίρι είναι η λύση μιας μακράς διαμάχης στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Γνωρίζουμε τις αντικσότητες, την εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση των ΙΠΑ σε σχέση με τα Airbus. Όμως το ψήφισμα δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα και θα προτείνουμε πολύ μικρές ε, αλλαγές στη διατύπωση και προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το παν για να καταλαγιάσει τις εντάσεις. Ευχαριστώ. Για τους πρασίνους παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καλό, πολύ καλό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσουν οι τόνοι και να διατηρηθεί πολυμερής προσέγγιση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Ήταν και το, το διάβημα Juncker το 2018. Πρέπει όμως να υπάρχει αμοιβαιότητα. Ποιε είναι οι δεσμεύσει των Αμερικανών. Ο πρόεδρος Τραμπ με την υπόθεση Airbus δείχνει τα αντίθετα. Το θυμήσατε κι εσείς, Πρόεδρε, όταν μιλήσατε στην Επιτροπή. Όταν μας κοινοποιεί ότι αποσύρει τη χώρα του από τη Συμφωνία των Παρισίων. Πώς κατευνάζει δηλαδή η Αμερικανική πλευρά τις εντάσεις και τις κατευνάζουμε μόνο εμείς αμοιβαία θα πρέπει να είναι η προσέγγιση. Οι, Ευρωπαίοι, η Γεωργοί είναι στο παριθώριο και το προ, στο προσκήνιο είναι τα γερμανικά συμφέροντα της γερμανικής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε, αλλά να καθυστερήσουμε τις διαβουλεύσεις για να σταλεί σαφές μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ. Να δείξει επιτέλους καλή θέληση και εκείνος από την πλευρά του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 να σας ευχαριστήσω και για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής και για την ετοιμότητα που έχετε να επιταχύνετε την εξέλιξη των πραγμάτων. Ελπίζω να εγκριθούν αυτά πριν το τέλος της χρονιάς. Δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο του ΕΛΚ. Είναι σημαντική συμφωνία και το είπατε κι εσείς με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να παραμείνουν, δηλαδή η ποσόστοση θα παραμείνει η ίδια, και δεν θα μπορούμε να εισάγουμε κρέας που ε, υφίσταται ορμόνες, έχει ορμονών και τα λοιπά. Και καλώς. Στην Αργεντινή όμως έχουμε ποσοστώσεις εκεί και δεν υπάρχει καμία αποζημίωση και κανένα αντιστάθμισμα. Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο φάκελος και μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε επικοδομητικό διάλογο με τη ΣΥΠΑ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν χάσει τη θέση που είχαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άρα να έρθουμε εμείς να ανισχύσουμε τη θέση μας εκεί και να ελπίζουμε ότι είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μην περιοριστούμε στο κοινοβουλευτικό διάλογο, αλλά στο ύψιστο επίπεδο πολιτικού διαλόγου με την ΣΥΠΑ να ε, τεθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, κύριε Σιγητά. Προφανώς όλα συνδέονται μεταξύ τους και όταν μιλάμε για εισαγωγές βόηου κρέατος και ποσοστώσεις, προφανώς και αυτό σχετίζεται και με άλλα αγαθά και άλλα προϊόντα. Ε, ανεξάρτητα από αυτό, ε, οι εισαγωγές ε, κρέατος έχουν άμεση σχέση και με την κλιματική αλλαγή αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να περιοριστεί η κατανάλωση κρέατος. Έχω ένα ερώτημα, θεμελιώδες κατά την άποψή μου. Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι ποσοστώσεις, λόγω του ότι έχουμε άλλες χώρες που εξάγουν κρέας, οι ποσοστώσεις αυτές τις άλλες χώρες δεν έχουν αλλάξει. Γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει ότι λόγω της συμφωνίας Μερκοσούρ θα προσθεθούν ποσοστώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, ξεβρέτει μία λύση η οποία υποτίθεται ότι ε, λύνει το πρόβλημα ενός εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ ή τουλάχιστον το λύνει κατά τη Από τις ΗΠΑ βέβαια αυτή τη στιγμή ε, δεν έχουμε κάποιο αντάλλαγμα. Αυτό αναφέρεται στη γνωμοδότηση στο ότι όσον αφορά τους δεσμούς για το χάλιβα και το αλουμίνιο εκεί δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ας μην ξεχνάμε τι ακριβώς συμβαίνει και με το Airbus και το Boeing στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Όλα αυτά δημιουργούν ε, πρόβλημα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ε, με αυτή τη λύση του ΠΟΕ μπορεί να ξεβρεθεί κάποιο πρόβλημα, κάποια λύση. Ε, οι πράσινοι πράγματι έχουν μια διπλωματική στάση, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές θα πρέπει οι ΗΠΑ να αλλάξουν τη θέση τους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μορέλ, δεν θα προσθέσω πολλά στα λεγόμενα του κυρίου Σόλτς, όμως ακούω πάντοτε με μεγάλη προσοχή τα λεγόμενα του κυρίου Μπέρτ Λάγκε και λέτε, χαιρετίζει και αναγνωρίζει το γεγονός ότι παρόλο που είναι δύσκολο να ξέρει κανείς αν προβλέπεται αντιστάθμισμα ή αποζημίωση, τα λοιπά μέρη του ΠΟΕ και το καθεξής. Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν προβλέπεται αποσμίωση, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι προβλέπεται. Υπάρχει αυτή η συμφωνία και λέμε θαυμάσια με τι έχουμε. Η Αργεντινή, η Νέα Ζηλανδία δέχονται να μειώσουν την ποσόστοση από 30.000, 33.000 στους 10.000 τόνους και ούτω καθεξής. Υπάρχει το project με Mercosur και το project με την Αυστραλία. Πιστεύετε πραγματικά ότι η Αυστραλία πρόκειται να υπογράψει μια συμφωνία ελευθέρου ε, εμπορίου που να μειώνει την ποσόστοσή τη. Με πονηριά μπαίνει αυτή η πρόταση. Εμεί γνωρίζουμε όμω την απάντηση. Ποτέ δεν θα το πράξει. Λέμε χωρίς ορμόνες. Ναι, αλλά προέρχονται από αγροκτήματα και κτηνοτροφικά κέντρα με 10.000 βοηθοί μέσα, τα οποία τα παχαίνουν με, γιατί τα μπουστάρουν με αντιβιωτικά. Είναι πολύ βιομηχανική παραγωγή κρέατος αυτή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεσέγλο. Ντεσέγλο. Όχι Ντεκέρλε, πρόεδρε, που με λέτε. Ντεσέγλο. Θέλω να στηρίξω τους προλαλήσαντες. Νομίζω ότι τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να διευκολύνουμε τη συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι εννοώ όμως. Ο κτηνοτρόφος, βοηού κρέατος, στο αγρόκτημά του, δυσκολεύεται να καταλάβει όλα αυτά τα οποία λέμε εμείς εδώ. Και υπάρχει αυτή η πίεση από τις ε, ε, επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου που ζητούν να πάρουν κάποιο αντιστάθμισμα, κάποιες εγγυήσεις, κάποιες εξασφαλίσεις και ευλόγως. Είναι χρήσιμο λοιπόν να αξιοποιήσουμε το πυρήνα της δουλειά σας, όμως να επιφέρουμε κάποιες εγγυήσεις, κάποιες ε, διαβεβαιώσεις στον κλάδο. Νομίζω ότι και στη δική μας Επιτροπή και στη Γεωργική Επιτροπή αυτό που προκύπτει συνέχεια όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει διεθνή συμφωνία είναι ε, το βόλιο κρέας, το οποίο τίθεται ξανά και ξανά επιτάπητος. Άρα να χαιρόμαστε για το ότι έχει βελτιωθεί η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΕΠΑ, ΕΕ, αλλά να μην λησμονούμε ότι ο κλάδος του βόηου κρέατος θα πληγεί. Θα έχει άμεσο ή έμεσο αντίκτυπο από τις αποφάσεις μας. Να το προσέξουμε αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια έχω να κάνω. Το πρώτο για το, τις ορμόνες και τα αντιβιωτικά και τα feedlots, αυτά τα τεράστια αγροκτήματα. Κανένα προϊόν το οποίο δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί βόλιο κρέας το οποίο θα εξαχθεί στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτό το ποσοστό. Αναφερθήκατε στα feedlots, σε, αυτά, ε, σε αυτές τις γιγαντιές τα ίστρες αν θέλετε. Ε, δεν υπάρχουν μόνο στη ΣΥΠΑ ξέρετε, υπάρχουν και σε εμάς δεν θα καταλήξουμε να εισάγουμε περισσότερο βόλιο κρέας. Η προέλευση του θα μοιραστεί και θα κατακαιρματιστεί και θα διανεμηθεί αναλόγως με την πρόταση που, είναι, που βρίσκεται επιτάπητος. Τώρα, οι συνέπειε για την αγορά βοηού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει επιπρόσθετο βόλιο κρέας που θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτή την πρόταση. Αυτό που επιτρέπεται με αυτή την ποσόστοση ήδη μπαίνει στην Ένωση τα τελευταία χρόνια. Και σε σχέση με την, το αντιστάθμισμα, θέλω και εγώ να επιμείνω σε αυτό που είπα πριν. Δεν προβλέπεται αντισταθμίσματα, γίνονται διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, η διαπραγμάτευση έχει τη δική της δυναμική το εγχείρημα που έχουμε μπροστά μας σήμερα είναι ένα εγχείρημα με ισορροπία. Η μείωση στις ποσότητες που δίδονται σε ορισμένους προμηθευτές δεν θα δίνονται για να δοθεί αντιστάθμισμα κάπου αλλού. Το λέμε αυτό ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει αντιστάθμισμα. Είναι η ενεξελίξη διαπραγματεύσει, αλλά δεν υπάρχει δέσμευση και υποχρέωση να αντισταθμίσουμε με πρόσθετε ποσότητε κάπου αλλού. Αυτό δεν θα γίνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος και εγώ σα ευχαριστώ και ευχαριστώ και τα μέλη για τα σχόλιά τους. Βεβαίως δεν υπάρχει εγγύηση ότι επειδή δίνουμε αυτή την υποχώρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες θα προοδεύσουν οι σχέσεις μας. Θα το δούμε αυτό. Στις 13 Νοεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα. Θα ληφθεί απόφαση για τα ανταλλακτικά, για τα αυτοκίνητα και το καθεξής. Ε, είναι όλα αυτά κρεμή έχουν τάσει οι Ηνωμένε Πολιτείε να τα ανακατεύουν όλα, να τα βάζουν στο ίδιο καλάθι, το βόλιο κρέα με τα ανταλλακτικά, τα αυτοκίνητα και το καθεξή. Θα δούμε πώ θα ε, διαμορφωθούν οι εξελίξει. Νομίζω όμω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να δημοσιεύσουμε τη θέση μας και να την καταστήσουμε σαφή δημοσίως. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, η 10η Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 25 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα. Και με αυτά ολοκληρώνουμε την εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και μπαίνουμε τώρα στην εξέταση του σημείου, ξεκινούμε την εξέταση του σημείου 19 της ημερήσιας διάταξης, προσχώρηση ε, για τα νησιά Σολομώντα στην Συμφωνία Ενδιάμεσης Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών του Ειρηνικού Ωκεανού. Λάβαμε το αίτημα να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ε, για αυτή την προσχώρηση για τα νησιά ε, Σολομώντα για την Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και νησιών του Ειρηνικού Τρεις είναι οι χώρες, τα νησιά Φίτζι, Παπούα, Νέα Γουινέα και τα νησιά Σαμόα. Και εμείς έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας για αυτές τις τρεις χώρες το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Επίτροπο, την Εμπορική Επίτροπο από τα νησιά Σολομόντα, την οποία και καλωσορίζω θερμά. Καλωσορίσατε. Και πριν σας δώσω το λόγο, τον Επίτροπο, με συγχωρείτε, θέλω να ακούσω την Επιτροπή σε Πιγιό, η οποία θα μας παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλησπέρα ε, στους, στον εισηγητή Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω λιγάκι για την προσχώρηση άλλη μιας χώρα του ειρηνικού στην ε, Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ε, με τον ειρηνικό. Παλαιότερα είχαμε 14, τώρα έχουμε άλλε τρει, Έχουμε τρεις που ε, αποτελούν μέρος συμφωνία. Φίτζι, Παπούανα, Γουινέα και τα νησιά του Σολομόντα προσθέθηκαν πέρσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περιοχή πολλέ χώρε του ειρηνικού επιθυμούν να προσχωρήσουν σε αυτή την συμφωνία. Και σήμερα λοιπόν εξετάζουμε την προσχώρηση των, των νήσων του Σολομόντα. Η Υπάρχουν, όπως σας είπα, αρκετές χώρες του ειρηνικού. Ε, ο Τόγκα, η Λαρούσα, αυτές έπονται. Δεν είναι μία νέα συμφωνία, αλλά είναι μία συμφωνία που ήδη υπάρχει ε, και θα ε, διαφέρει θα προσφέρουμε ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά μας σε αυτές τις χώρες του ελληνικού ε, γιατί αυτές, τις, αυτές οι χώρες ε, χρειάζονται κάποιες ε, εγγύησει για ελεύθερη πρόσβαση. Αυτό ισχύει και για τα νησιά του Σολομόντα. πέρα όμως από το ότι δίνουμε ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά μας, υπάρχουν και συμφωνίες αμοιβαιότητας με ασύμετρο όμως τρόπο. τα νησιά του Σολομόντα δεσμεύονται να μειώσουν δασμούς από προϊόντα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι ε, οικοδομικά υλικά ε, κυρίως και η αγορά θα ανοίξει όλο και περισσότερο σε διάρκεια 15 ετών. Αυτό εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συμφωνία που έχουμε με τα νησιά του Ειρηνικού. Αυτά είναι μακριά βέβαια και από πλευρά πληθυσμού ε, δεν είναι και πολύ σημαντικά, δεν είναι πολύ σημαντικές ε, οι εμπορικές ε, ροές. Μιλάμε για 0,1% του ε, συνολικού εμπορίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς αυτό είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά για εκείνες τις χώρες όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, κυρίως για την αλία. Και αυτό ισχύει κυρίως για τα νησιά του Σολομόντα, ε, οι εξαγωγές τους ε, είναι καθοριστικές για τη χώρα αυτή, ε, δημιουργούν θέσεις ε, απασχόλησης και προσφέρουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό που έχει πει συμφωνία, έχει σημασία με αυτή τη συμφωνία, είναι ότι η περιοχή έχει γεωστρατηγική σημασία. Ε, με τις ε, εταιρικέ μας σχέσεις ε, με αυτά τα νησιά φτάνουμε σε ένα άλλο επίπεδο σχέσεων, προκύπτει διάλογος και προκύπτουν και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτά είναι θέματα που φαντάζομαι όσοι από εσάς έχετε δει τις συμφωνίες σε λεπτομερή βάση θα έχετε διαπιστώσει ότι ε, δεν υπάρχει εκεί ένα ολόκληρο κεφάλαιο ε, για την ανάπτυξη. Υπάρχει ένα άρθρο, βασίζεται στην αρχή της Συμφωνίας ε, του Κοτονού και αυτό είναι σημαντικό, αλλά σας λέω, δεν υπάρχουν αυτά τα κεφάλαια που βλέπουμε σε άλλες συμφωνίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς ε, χρησιμοποιούμε αυτή τη συμφωνία για να δείξουμε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, παρότι βιώσιμη ανάπτυξη δεν υπάρχει κατ' ουσίαν σε αυτή τη συμφωνία. Παράδειγμα, η τελευταία αποστολή έγινε τον Οκτώβρη στα νησιά Φίτζη και εκεί έγινε εκτενή συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι δύο πλευρές ε, δεσμεύτηκαν να ε, συνυπογράψουν μία σύσταση για τη βιώσιμη ανάπτυξη υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν και τις δύο πλευρές και εκεί ε, θέλουμε να συνεχιστούν οι συζητήσεις, το χάρη κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέματα βιοποικιλότητας ε, αποψήλωσης, ε, διαχείριση αλλιευτικών πόρων. Αυτά είναι θέματα όπου μπορούν να υπάρξουν ε, περαιτέρω συζητήσεις και όπου μπορούμε να προάγουμε τις αρχές μας. Όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, κατ' ουσίαν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή που να προβλέπεται στη συμφωνία, αλλά χρησιμοποιούμε την ευκαιρία που μας δίνει η συνεργασία για να συμπεριληφθεί η κοινωνία των πολιτών ε, στις εξελίξεις ε, ε, στο Φίτζι οργανώσαμε μία συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών. Είχαμε περίπου 100 ε, ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν ε, σε αυτή τη συνάντηση. Είχαμε εκπροσώπους επιχειρήσεων, συνδικάτων, ΜΚΟ. Όλοι αυτοί ήρθαν για να συζητήσουμε και για το τι μπορεί να προκύψει. Άρα δηλαδή όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και επίση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά δεν γράφονται αναλυτικά στη συμφωνία. Ένα άλλο θέμα που θέλω επίσης να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η συμφωνία έχει και μια ουσιαστική περιφερειακή διάσταση. Δεν είναι δηλαδή απλά μια συμφωνία ανάμεσα σε εμά και τα νησιά του Σολομόντα. Είναι μια συμφωνία που προάγει ε, το εμπόριο ανάμεσα ε, σε εμά και στις χώρες του Ειρηνικού, που βέβαια είναι πολύ μικρές σε διάσταση και δεν μπορούν αυτόματα να αναπτυχθούν σε πολλούς τομείς. Πρέπει να ε, στόχο πρέπει να έχουν και να μπορούν να αναπτύξουν οικονομίες κλίμακας ε, για την παραγωγή. Άρα δηλαδή οι συμφωνίες αυτές ε, καθορίζουν ένα πλαίσιο για να γίνουν συζητήσεις περί εμπορίου. Και σας είπα ότι ε, προκύπτει περιφερειακό εμπόριο και περιφερειακή αλυσίδα αξίας. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο της έκθεσης. Η σχέση με, τις υπερπόντιες, ε, με τα υπερπόντια διαμερίσματα, Νέα Καλλιδονία, Γαλλική Πολυνησία, η σχέση με αυτά τα διαμερίσματα είναι σημαντική γιατί και αυτά εντάσσονται στην περιοχή και έχουν καλές σχέσεις με τις χώρες του ειρηνικού. Ε, εδώ η εταιρική ε, συμφωνία θέλει να συμπεριλάβει καλύτερα αυτά τα διαμερίσματα ε, στον σύμπλεγμα των νησιών του ειρηνικού. Άρα δηλαδή μας ενδιαφέρει και η σχέση με τις υπερπόντιες εκτάσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτή την έκθεση. Ο κύριος Ράνχολ Πρένα, επικεφαλής της ε, αρμόδιας διεύθυνσης, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Νομίζω δεν είναι εδώ. Και ως εκ τούτου θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο Εμπορίου των Ισιών Σολομώντα για πέντε λεπτά. Στον, με συγχωρείτε, είναι κύριος, ο Επίτροπος του Εμπορίου. Ε, αγαπητά μέλη αυτής της ε, Επιτροπής, καταρχήν ε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνω μια σύντομη παρέμβαση ε, σχετικά με την επιδίωξη των νησιών του Σολομώντα να προσχωρήσουν ε, σε αυτή τη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παππούα, Νέα Γουνέα, Φίτζι και Σαμόα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για αυτή την εμπεριστατωμένη έκθεση επί του θέματος. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομόντα αντιμετωπίζουν το εμπόριο ως ένα καθοριστικό στοιχείο, ως ένα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, στόχοι του 2030. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομώντα είναι πεπισμένα ότι με την προσχώρησή μας και με τη συμμετοχή μας στην ενδιάμεση συμφωνία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο ως ένα εργαλείο το οποίο ε, θα προσφέρει δυνατότητες για να επιδιώξουμε την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη μείωση της φτώχειας. Θα μας επιτρέψει επίσης η συμφωνία να αντιμετωπίσουμε και άλλες ε, ε, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία μας. Ε, μας ενδιαφέρει να προσχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Κάτι τέτοιο αναμφίβολα θα βοηθήσει τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε τη διαφοροποίηση της παραγωγής να διευρύνουμε την περιορισμένη οικονομική μας βάση, θα μας βοηθήσει αυτή η συμφωνία να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις. Ως οικονομία ενός μικρού νησιού, αγωνιζόμαστε να ενταχθούμε στο ε, σύστημα του πολυμερούς εμπορίου και συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες ε, που έχουν σχέση με, τον, με τη μονομέρεια και τον προστατευτισμό ε, που αντιμάχονται τα συλλογικά συμφέροντα του πλανήτη. Ε, αυτή η συμφωνία θα συνεπάγεται καλύτερες ευκαιρίες για τις γυναίκες, ε, τα παιδιά, ε, για τους απόκληρους της κοινωνίας να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οικονομικής ανάπτυξης και με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, τρόφιμα, ασφάλεια με ε, τη συνεργασία μας με άλλες χώρες του ειρηνικού στο πλαίσιο του ε, αφηγήματος του μπλε ειρηνικού που εγκρίθηκε από τον ε, εκπρόσωπο της ΣΑΜΟΑ θα τορθώσαμε να επιτύχουμε συνεργασία σε θέματα αλλία, κλιματικής αλληγής, διαχείρισης των ωκεανών, ασφάλεια. Μπορέσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε οικονομικές ευκαιρίες, ευκαιρίες οι οποίες ε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομόντα επικύρωσαν τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και κατόπιν τούτου ε, τα νησιά του Σολομόντα επιθυμούν να εισάγουν την τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Παράδειγμα, η κυβέρνηση ε, κατασκευάζει μία υδροηλεκτρική μονάδα για να αντικαταστήσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων ε, για την ε, παραγωγή ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι εταίροι μας μας στηρίζουν με επενδύσεις ε, για την ηλιακή ενέργεια, για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, αυτά στα σχολεία μας, στην τοπική κοινωνία. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι αποφασισμένη να περιορίσει τις εκπομπές μας κατά 50% μέχρι το 2050. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομόντα έχουν ολοκληρώσει τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της αλίας και τώρα έχουμε ένα από τα καλύτερα καθεστώτα διαχείρισης αλίας στον ειρηνικό. Με την ε, νομοθετική πράξη ε, διαχείρισης αλίας του 2017 έχουμε μηχανισμούς εντοπισμού αλλιευτικών προϊόντων και μπορούμε έτσι να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται με τα ψάρια μας από την ώρα που ε, γίνεται η περισυλλογή τους μέχρι τις εξαγωγές, την, ε, την εξαγωγή στις ε, ευρωπαϊκές αγορές. Ο τομέας της αλίας για μας είναι καθοριστικός. Καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών του Σολομόντα, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ασφάλεια τροφίμων της χώρας η μόνη μονάδα επεξεργασίας ε, τόνου ε, στο νησί ε, απασχολεί 77 γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και εμείς να προσχωρήσουμε σε αυτήν την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέσης έτσι ώστε να αποκτήσουμε δυνατότητες εξαγωγών συμπεριλαμβανομένων και των αλλιευτικών προϊόντων. Κύριε Πρόεδρε, το 2018 Είχαμε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και εκεί ε, συστήνεται στα νησιά της Σολομόντα από ε, καθεστώς ε, λιγότερο αναπτυγμένης χώρας να περάσει σε μία ανώτερη βαθμίδα μέχρι το 2024. Γι' αυτό τα νησιά της Σολομόντα πλέον ε, επεξεργάζονται μία στρατηγική η οποία αναγνωρίζει ότι το εμπόριο είναι ένα βασικό εργαλείο που θα διευκολύνει την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Τα νησιά του Σολομόντα θα χαράξουν ε, ένα βιώσιμο μονοπάτι που θα μας ε, επιτρέψει να περάσουμε σε άλλη φάση αυτό βέβαια θα βοηθήσει και στην ε, δημογραφική έρευνα που θα γίνει από τα ε, μέσα Νοεμβρίου μέχρι και την επόμενη χρονιά. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομόντα έχουν ένα μηχανισμό που επιτρέπει σε, στην κοινωνία των πολιτών ε, σε, στον ιδιωτικό φορέα να συμμετέχουν στην χάραξη της εμπορικής πολιτικής. Έχουμε το Συμβούλιο, Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξη Εμπορίου, NTDC είναι το κρονίμιό του, που μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε η ανάπτυξη να είναι ολιστική, χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων. Ε, αυτού του Συμβουλίου προείσταται ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου, που είναι επίσης και ο Υπουργός που έχει και το χαρτοφυλάκιο για το εξωτερικό εμπόριο. Μέσω αυτού του Συμβουλίου έχουμε μπορέσει να συμμετάσχουμε σε διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες με άλλους εταίρους. Προφανώς ε, οι διαπραγματεύσεις αυτές αφορούν και αυτή την ενδιάμεση συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική που αναφέρεται στην έκθεση του εισηγητή περιλαμβάνει και τα γεωπολιτικά θέματα που αφορούν στα νησιά του Σολομόντα. Πρόσφατα συνήψαμε διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω εσάς, τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, ότι οι τελευταίες αποφάσεις ε, που λάβαμε ε, για να συστήσουμε διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν στο πνεύμα της εκπλήρωσης ε, των υποχρεώσεών μας ε, για να εφαρμόσουμε το ψήφισμα 2758 κάθετος 71. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα δίνει τότε δυνατότητα στα νησιά της Ολομόντα να ενταχθούν και αυτά στη μεγάλη οικογένεια, στην πλειοψηφία των κρατών των Ηνωμένων Εθνών, συμμελωμένες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δέχονται το ψήφισμα. Όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα, να σας ε, διαβεβαιώσω ότι είμαστε μια νεόκοπη, ε, φιλόδοξη δημοκρατία, ε, εφαρμόζουμε διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση των νησιών του Σολομόντα αναγνωρίζει τη σημασία των δασών και η κυβέρνησή μας για το λόγο αυτό έχει λάβει και μέτρα για να αντιμετωπιστεί η παράνομη λοτομία η κυβέρνηση είχε αναθεωρήσει την τις νομοθετικές πράξεις για, την, ε, για τα δάση. Ε, θέλουμε να διαχειριζόμαστε τα, τα δάση με, με βιώσιμο τρόπο μέχρι και το 2020. Και έτσι η κυβέρνηση θα ρίνει επενδύσεις ε, μεγάλης κλίμακας στην, στις πολιτικές αναδάσωσης Επίσης, ε, η κυβέρνηση ενθαρρύνει διαδικασίες προς τα κάτω. Επίσης, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ε, χρησιμοποιήσει την λογική εκμετάλλευση της δασοκομείας ε, μέχρι το 2023. Θέλουμε να προσχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία για να ενισχύσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τις υπερπόντιες χώρες στον ειρηνικό. Και αυτό σημαίνει μέτρα όπως χρήση παραγωγής με βάση την αλυσίδα αξίας. Τα νησιά του Σομολόντα επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτές τις συμφωνίες και η Πολυνησία και η Νέα Καλλιδονία. Αυτή είναι μια τάση που δεσμευόμεθα να την διαφυλάξουμε και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν να είστε σίγουροι ότι τα νησιά του ε, Σολομώντα θα συνεργαστούν επικοδομητικά με τα υπερπόντια διαμερίσματα. Κύριε Πρόεδρε, τα νησιά του Σολομόντα... Ε, προσπαθούν ε, να ε, εφαρμόσουν και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες που εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Παππούα Νέγου Νέα, η Σαμό και τα νησιά Φίτζη θέλουν, θέλουμε να συνεργαστούν μαζί μας για να είναι η περιοχή πιο σταθερή και για να έχουμε καλύτερες εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη. Να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τις ε, ευκαιρίες ε, που ε, προσφέρονται από τις συμφωνίες, γιατί στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε, να σας απευθύνω το λόγο για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις ολοκληρωμένες σας ε, και περιστατωμένες εξηγήσεις για την ε, εμπορική κατάσταση αλλά και τη γεωπολιτική κατάσταση στα νησιά Σολομώντα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Και σας ευχαριστούμε που κάνατε αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι από τα νησιά Σολομώντα στις Βρυξέλλες. Μόνο και μόνο για αυτή τη σημερινή μας συμμενεδρία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στρέφομαι, στρέφομαι στην εισηγήτρια, την κυρία Ζαμή. Έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αντικαθιστώ τον κύριο Ρουζέ ο οποίο δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα παρουσιάσω λοιπόν την έκθεση εξ ονοματό του. Και θα ξεκινήσω με τρία νούμερα. Το 2018 από τα νησιά του Σολομόντα είχαμε από το εξωτικό ξύλο, από κονσέρβες ε, ψαριού και από ε, φινικέλαιο τις εξαγωγές. Τρεις ε, τομείς, τρία προβλήματα. Είναι λίγες ίσως οι ποσότητες, ναι μεν, αλλά θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο την εκτίμησή μας να την βασίσουμε στις γεωπολιτικές και περιβαλλοντικές πολιτικές πτυχές για μια ενδεχόμενη προσχώρηση των νήσων Σολομόντος σε αυτή τη συμφωνία. Ναι, πράγματι τα νησιά του Σολομόντα βρίσκονται σε μια στρατηγική περιοχή από πλευράς βιοπικιλότητας και σίγουρα είναι ένας φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νήση Σολομόντος. Όμως, η νήση Σολομόντος και το είπε και ο υπουργό. Πρόσφατα έχουν προβεί σε διπλωματική προσέγγιση με την Κίνα. Δικαίωμά του βέβαια ε, υπέγραψαν πολλές συμφωνίες διμερείς δε. Και η κινέζικη στήριξη στις υποδομές των ίσων Σολομόντος ε, θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιες εξελίξεις που δεν μπορούμε να μετρήσουμε ακόμη τι αντίκτυπο θα έχουν και τι να θα, θα υπάρξουν. Και έρχομαι στην αλία. Όλοι γνωρίζουμε ότι συχνά χωρίς έγκριση αλλιεύουν τα κινέζικα πλοία κοντά στις ακτές του Νότιου Ειρηνικού, στα χωρικά, κοντά στα γαλλικά χωρικά ύδατα. Και πρέπει να σας πω, στο συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αλλά συχνά, πώς να το πω, δεν υπάρχει επαρκή επιτήρηση από τι τοπικέ αρχέ ε, των νήσων Σολομόντο ω προς αυτό και όλα αυτά φυσικά έχουν περιβαλλοντικέ επιπτώσει. Η Κομισιό δεν μπορεί να τι αρνηθεί. Επίσης να προσθέσω ότι η Κίνα, μην το ε, ξεχνάμε αυτό, ε, θα εποφεληθεί από τι υποδομέ εκεί και σε ό,τι αφορά την προσχώρηση των νησών Σολομόντων σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία εταιρική σχέση, τελικά την κινέζικη βιομηχανία θα ωφελήσει. πάντοτε μιλώ για την αλία. Επομένως, από την πλευρά μας ε, επιφυλάξεις έχουμε να εκφράσουμε για τα οικονομικά και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που γνωρίζουμε ότι ε, σε αυτά είναι προσιλωμένοι. Δεύτερον, για το εξωτικό ξύλο το οποίο προέρχεται από τις νήσεις Σολομόντος. Συνήθως ε, προς την Κίνα γίνονται εξαγωγές τέτοιων προϊόντων αν προσχωρήσει στην διάμεση συμφωνία όμω, θα υπάρξουν νέε διάβλοι και διέξοδοι προ τι ευρωπαϊκέ αγορέ. Νομίζω ότι αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση, για να μην πω θα καταστρέψει ε, τα δάση του αρχιπελάγου. Να σας υπενθυμίσω, ε, επειδή στην τελευταία θητεία είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τη συμφωνία του Βιετνάμ. Και εκεί λάβαμε την προφύλαξη να προσθέσουμε ένα πρόσθετο ακριβώς κείμενο το οποίο εμποδίζει τη διακίνηση, την εμπορία παράνομου, παράνομης ξυλίας. Οι εξαγωγές τώρα λέω δεν είναι σημαντικές σε ποσότητες, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία που θα αυξήσει έστω και ε, περιθωριακά ε, τις εξαγωγές ε, λέω στην Ένωση, εφόσον εξανιστάμεθα με αυτό το θέμα γενικώ. Πώς θα ψηφίσουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Και τέταρτον να πω το είχα πει και νωρίτερα. Ε, συζητήσαμε και τη συμφωνία με τη Σαμόα, τη Σαμόα. Εμείς θέλουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας, ε, όχι τα γαλλικά μόνο, αλλά και τα ενωσιακά, τα ευρωπαϊκά. Επομένως τα ίδια αίτια έχουν τα ίδια αποτελέσματα, πρέπει να το έχουν υπόψη. Δεν θέλουμε εδώ ε, να επιβάλλουμε έναν κακώς εννοούμενο προστατευτισμό. Απλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαίο όφελος από όλες τις πλευρές. Και βέβαια και το περιβάλλον πρέπει να έχουμε κατά νου. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι εμείς θα απορρίψουμε αυτή την συμφωνία. Ευχαριστώ. Κριστόφ Χάνσεν αντί του Ντάβιντ Μακάλιστερ. Θα τα πείτε γερμανικά τώρα δηλαδή, γιατί έχετε μιλήσει όλες τις γλώσσες. Όχι. Αγγλικά θα τα πω και αυτή τη φορά, γιατί τα λέω και πιο γρήγορα και θα δουλέψουν λιγότερο οι διερμηνείς, λέει ο κύριος Χάνσεν. Υποστηρίζει το ΕΛΚΑ την προσχώρηση των ίσων Σολομόντων στην διάμεση συμφωνητερική σχέση ε, για πέντε βασικού λόγου. Ε, την παρουσία ενός ακόμη κράτος του ειρηνικού που θα δώσει περισσότερη δυναμική ε, σε αυτή τη συμφωνία, ε, κάτι το οποίο συνάδει με την προσέγγιση της Κομισιόν Δεύτερον. Η ενδιάμεση συμφωνία θα ενισχύσει την παρουσία της Ένωσης στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή όπου κυριαρχούν οι σχέσεις με την γειτονική Κίνα. Μπορεί να μην μπορέσουμε να επαναξισορροπήσουμε αυτές τις σχέσεις, όμως είναι σημαντικό να δώσουμε μήνυμα ότι μας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή και ελπίζουμε οι νέοι να το εκτιμήσουν. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνούμε με τα επιχειρήματα του εισηγητού. Τρίτον, η προσχώρηση των ίσων Σολομόντο θα δημιουργήσει ένα ε, ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού με άλλου εταίρου, του εταίρου που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Γιατί να αποτρέψουμε να έχει και η χώρα αυτή τα ίδια πλεονεκτήματα. Επίσης, ε, μπορεί να μην έχουμε ακόμη μεγάλες ε, επιπτώσεις ως άμεση συνέπεια αυτής της προσχώρησης, γιατί είναι ε, μικρής κλίμακας οι συναλλαγές και οι σχέσεις μας. Άρα και εδώ δεν συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία του συγητού ότι θα υπάρξουν τεράστιες εξαγωγές ποινικελαίου και εξωτικού ξύλου. Οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά πρέπει να εφαρμόζουν τις φυτογειονομικές διατάξεις, περιβαλλοντικές διατάξεις κτλ. Και η Κομισιόν θα παρακολουθεί εκ του σε αυτή τη συμφωνία και θα φροντίσει να μην ε, οδηγήσει σε απερίμωση ε, και ε, μάλλον σε αποψήλωση των δασών εκεί. Όπως και σε άλλες εμπορικές συμφωνίες, έτσι και εδώ θεωρούμε ότι η προσχώρηση των ίσων στην διάμεση συμφωνία είναι θετική και θα έχει ως αποτέλεσμα την πολύ καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών και στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα νησιά του Σολομόντα και η γενικότερη περιοχή του Ειρηνικού. Είναι πολύτιμη σύμμαχη τη Ένωση, ιδίω στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Για όλου αυτού του λόγου, η ομάδα του ΕΛΚ στηρίζει την προσχώρηση των Ισοσαλωμόντων στην διάμεση Συμφωνία Εταιρική Σχέση και θα προτείνουμε μια τροπολογία. Ε, δηλαδή, να μην γίνει δεκτή η πρόταση του εισηγητού, να μην γίνει δεκτή η προσχώρηση. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η εισηγήτρια δεν δέχεται την πρόταση για λόγους πολιτικούς και για λόγους του περιβάλλοντος αλλά εγώ νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δώσουν δυνατότητα στα νησιά του Σαλομόντα να ενταχθούν σε μια ε, σε ένα σύστημα, σε μια ε, τάξη πραγμάτων και έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τους περαιτέρω κινδύνους. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των 550.000 κατοίκων. Τόσοι είναι, αν δεν απατώμε. Τα νησιά του Σολομόντα είναι μια χώρα που δεν είναι ανεπτυγμένη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα δασμολογικών προτιμήσεων. Και πιστεύω ότι αυτή είναι και η καλύτερη λύση. Για μας, για τη δική μας πολιτική ομάδα, αυτή είναι η καλύτερη λύση. Βέβαια, ε, θα πρέπει μέσω της συμφωνίας να μεριμνήσουμε και για την ε, τήρηση των ε, διατάξεων. Και όλα αυτά μπορούμε να τα ελέγχουμε. Η δική μας η πολιτική ομάδα συμφωνεί με αυτή την πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκίψον, για το Renew. Ευχαριστώ. Δυστυχώς η σκιώδης συγγήτρια δεν είναι εδώ. Ε, δεν είναι εδώ ο εισηγητής και θέλω να παραθέσω τα λόγια του. Δεν συμφωνούμε με την τεκμηρίωση του εισηγητή, του κυρίου Αντρέ Ρουζέ, για τους εξής λόγους. Η οικονομική συμφωνία εταιρική σχέση με τις χώρες του ειρηνικού είναι κάτι που ήδη υπάρχει. Εδώ δεν ασχολούμαστε με νέα συμφωνία, αλλά με την πρόσβαση μίας χώρας σε μια συμφωνία που έχει ήδη υπογράψει και εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ανοίξουν νέες αγορές και δεν θα τεθούν σε κίνδυνο εδάφη είναι μια συμφωνία που συμφέρει κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει ελεύθερη πρόσβαση στα προϊόντα των χωρών του Ειρηνικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν θα είχαν και προτιμησιακό καθεστώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μπορεί να είναι περιορισμένες οι εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 51 εκατομμύρια ευρώ μόνο το 2019, είναι όμως πολύ σημαντικά για την οικονομία μιας τόσο μικρής χώρας, όπως είναι τα νησιά Σολομόντα. Έτσι γίνεται διαφοροποίηση του, της παραγωγής τους και αναπτύσσουν το δυναμικό τους. Αυτή τη στιγμή κάνουν μόνο εξορεκτική βιομηχανία και υλοτομία και μπορούν να διαφοροποιηθούν, να κάνουν γεωργία, να κάνουν αλληλεία. Και έτσι με αυτή τη συμφωνία θα αναπτυχθούν ουσιαστικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για μας και για αυτούς. Τα νησιά Σολομώντα και η περιοχή του Ειρηνικού ήταν πολύτιμη σύμμαχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκαθεν και ειδικά σε αυτόν τον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι μια χώρα αυλαβής, μικρή, νησιωτική, δεν, βρίσκεται στον κατάλογο του IUU της λαθρέας άναρχης και παράνομης αλίας, δεν βρίσκεται στον κατάλογο των χωρών που δεν είναι συνεργάσιμες φορολογικά δεν θα οδηγήσει αυτή η συμφωνία στην αύξηση των εξαγωγών της Κίνας και την αύξηση της επιρροής της Κίνας. Αντίθετα, θα αγκιστρωθούμε εμείς ως στέρεος οικονομικός εταίρος σε μια περιοχή την οποία, στην οποία κυριαρχούν άλλοι παίκτες και άλλοι παράγοντες, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία. Η συμφωνία αυτή δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη αποψήλωση των δασών και σε μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αντιθέτω, δίνει εργαλεία να υπάρξει δέσμευση από αυτέ τι χώρε και από τα νησιά Σολομόντα και από τις τρεις λοιπές χώρες. Επομένως, στηρίζουμε στεναρά την προσχώρηση των νησιών Σολομώντα σε μια ε, συμφωνία η οποία ήδη αποδεικνύεται επωφελής και για μας και για τις γειτονικές της χώρες, την Παπούα Νέα Γουινέα, τα νησιά Φίτζη και τα νησιά Σαμόα. Η Σεσίλα, από την Επιτροπή, παρακαλώ να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω κατά κύριο λόγο στο ερώτημα του εισηγητή στο θέμα, στα τρία συγκεκριμένα θέματα του εισηγητή και θέλω να υπενθυμίσω αυτά τα οποία μόλις μας ε, τόνισε η κυρία Γκίψον. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία της οικονομικής εταιρικής σχέσης για τη διαφοροποίηση της οικονομίας των νησιών Σολομώντα. Είναι αληθές ότι προς το παρόν και οι εξαγωγές και η παραγωγή των νησιών Σολομώντα περιορίζονται σε πολύ λίγους τομείς και κλάδους, αλλά σε μια οικονομική εταιρική σχέση ακριβώς αυτό το ρόλο διαδραματίζουμε. Βοηθούμε ε, για αυτή τη διαφοροποίηση, αναπτύσσουμε διάφορους κλάδους στη χώρα οικονομικούς, η κλάδη της ε, ε, γεωργίας είναι κλάδη προτεραιότητας, αλλά και κλάδη που έχουν να κάνουν με τον τριτογενή τομέα και τις υπηρεσίες και το καθεξής. Ε, όλα εξαρτάται από το κατά πόσο θα διαφοροποιηθεί η οικονομία τελικά, αλλά ε, παρόλο που η συμφωνία δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, σίγουρα θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφοροποίησης ε, της ε, οικονομίας της χώρας αυτής. Πιο συγκεκριμένα για το θέμα της αλληλεία για να διευκρινίσω, θέλω να πω τα εξής. Η συμφωνία δεν θα δώσει πρόσβαση σε αυτή την περιβόητη δυνατότητα του global sourcing, δηλαδή να επιτρέψουμε σε σκάφη αλλιευτικά που δεν είναι από τον Ειρηνικό ή από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελιεύσουν ψάρια και να γίνεται η επεξεργασία στα νησιά Σολομώντα και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμολογική επιβάρηση, χωρίς ποσοστός, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Μόνο η Παπούα Νέα Γουινέα είναι δικαιούχου αυτού. Ανταποκρίνεται σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και εγγυήσει. Και γίνεται πολύ σημαντική παρακολούθηση και εποπτεία της ε, χώρας αυτής για να έχει δικαίωμα σε ένα τέτοιο μέτρο. Δεν είναι κάτι που θα γίνει αυτόματα για τα νησιά Σολομόντα, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικά, σχετικό αίτημα και θα το εξετάσουμε ενδελεχώς και επισταμένως. Δεν θα μπορούν αλλιευτικά σκάφη που δεν ανήκουν στα νησιά Σολομόντα να αλλιεύουν ελεύθερα και να κάνουν ε, την επεξεργασία στα νησιά Σολομόντα και να εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανένα θέμα. Υπάρχουν πολύ δεσμευτικά μέτρα ε, και στο θέμα της αηφόρου ανάπτυξης για να ε, μπορεί η χώρα αυτή ε, να επωφεληθεί από το, τη χορήγηση καθεστώτος δασμολογικών προτιμήσεων. Ως προς την παράνομη υλοτομία, να σας πω ότι δεν εισάγουμε ξυλία από τα νησιά Σολομόντα αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, πρέπει να τεθεί είναι αληθινή η υπόθεση της αποψήλωσης των δασών. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει και στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης αλλά και στο επίπεδο των πολιτικών συζητήσεων μεταξύ Δουσιών ε, ε, Σολομώντα και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως εμείς δεν εισάγουμε ούτε θα εισάγουμε ξυλία, ε, πόσο μάλλον λαθρέα και παράνομη. Τώρα για το φινικέλαιο, σωστά τα λέει και ο εισηγητής, οι εισαγωγέ από την Ένωση προ τα νησιά Σολομόντα είναι πολύ μικρέ, περίπου 2% των εισαγωγών μα στο σύνολο για το φινικέλαιο. δεν είναι το θέμα να είναι κανείς υπέρ ή κατά του φοινικέλεου. Είναι το θέμα κατά πόσο παράγεται με βιώσιμο, με αηφόρο τρόπο. Οι εισαγωγέ μας από τα νησιά Σολομώντα ανέρχονται στο 2% των συνολικών εισαγωγών φινικελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κριτήρια που επιβάλλουν τα νησιά Σολομώντα είναι πολύ συγκεκριμένα για την αηφορία κατά την παραγωγή του φινικελαίου. Πήγαμε εμεί στη χώρα αυτή ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήγαμε και τα είδαμε σε ε, την παραγωγή, η οποία γίνεται σε σωστέ συνθήκε. Τώρα, ε, θέλω αυτά για να απαντήσω στα συγκεκριμένα ερωτήματα, όμως η Επίτροπος και ο Πρέσβης είναι ε, καλύτερη, σε καλύτερη θέση για να εξηγήσουν τα πολιτικά της συμφωνίας και τους ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Αυτά για τα τεχνικά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για μια σύντομη παρέμβαση, ο κύριος Μπρέντερ, επικεφαλής του τμήματος ή της διεύθυνση για τις χώρες αυτές, για τον Ειρηνικό, την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις ευρύτερες προοπτικές και ένα ευρύτερο πολιτικό σκηνικό όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς Θεωρούμε ότι τα νησιά Σολομώντα είναι σημαντική εταίρη για εμάς και άλλες χώρες της περιοχής, προκειμένου να διατηρήσουμε τη διεθνή τάξη πραγμάτων η οποία βασίζεται σε κανόνες. Και τα νησιά Σολομώντα θέλουν να εμπλακούν σε μια δέσμευση μαζί μας, να δεσμευτούν μαζί μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και συνεργάζονται μαζί μας στα διάφορα πολυμερή φόρουμ και κυρίως στο πλαίσιο του ΑΕΕ όπως και άλλες γειτονικές τους χώρες, για να καταπολεμήσουμε από κοινού την κλιματική αλλαγή και αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι αναφέρθηκε το γεγονός ότι τον ειρηνικό αυτή τη στιγμή το να διεκδικούν διάφοροι παίκτες. Όντως πράγματι συμβαίνει αυτό και πιστεύουμε ότι η προσχώρηση σε μια οικονομική εταιρική σχέση θα αγκιστρώσει τα νησιά Σολομώντας περισσότερο και πιο στέρεα στη δική μας τροχιά, στη δική μας διαδρομή και αυτό θέλουμε να το δούμε, θέλουμε να φανεί και να ακουστεί και στη Καμπέρα ε, και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κάτι που έχει υποθεί προηγουμένως, ότι είναι μια πολύ φτωχή χώρα. Θέλω να το τονίσω και εγώ αυτό. Και θέλουμε ακριβώς με τη συνεργασία μας που περιλαμβάνει και αναπτυξιακό σκέλος, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ε, αυτού του νησιού. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις αρχές της νησιωτικής αυτής χώρας και, ε, και σε θέματα εμπορικά. Είναι προς όφελος όλων να προωθήσουμε την ανάπτυξη των νησιών Σολομώντα και αν κάτι είναι ατελές και δεν είναι πολύ καλό σήμερα, με καλή συνεργασία θα λυθεί. Θα λυθεί και διμερός και σε περιφερειακό επίπεδο. Άστα ε, ας προχωρήσουμε μαζί από κοινού και να λύνουμε τα προβλήματα κάθε φορά που προκύπτουν. Ευχαριστώ. Και για να ε, ολοκληρώσουμε η εκπρόσωπος του εισηγητή, η κυρία Ζαμέ, το λόγο. Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς εμένα. Είπα ότι ο όγκος των συναλλαγών μπορεί να είναι μειωμένος, όμως ο αντίκτυπος του είναι σημαντικός, σε επίπεδο γεωπολιτικό και περιβαλλοντικό. Θα σας θυμίσω και ε, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι σε καμία περίπτωση εδώ, όποιος και αν είναι, δεν έλαβε υπόψη του τον αναπόδραστο παράγοντα που ακούει στο όνομα Κίνα. Δεν λέω να μην κάνουμε δουλειέ με τα νησιά Σολομόντα, αλλά να διατηρήσουμε ο καθένα τα συμφέροντά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα συμφέροντά τη. Ε, παραμένω στη θέση μου. και για την αποψήλωση των δασών. Πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις και να υπάρχουν στο κείμενο. Εν τω μεταξύ με μεγάλη χαρά μαθαίνω ότι ε, τίθεται στο περιθώριο η προβληματική για το, ε, όλη αυτή η παρουσίαση των απόψεων για το φινικέλαιο. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνει η εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Εμπορίων των Ισιών Σολομώντα για την ε, ε, επίσκεψή του στην Επιτροπή μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 6 το απόγευμα 14 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου. Με αυτά ολοκληρώνουμε την εξέταση του σημείου 19 της ημερήσιας διάταξης. Ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 20 και χαίρομαι ιδιαίτερως διότι η Σεσίλια Μάλστρομ, αρμόδια επίτροπος για το εμπόριο, είναι εδώ μαζί μας. Ίσως είναι και η τελευταία φορά που μας επισκέπτεται στην Επιστροπή Ίντα. Αλλά βέβαια δεν είναι και βέβαιο αυτό, κανείς δεν ξέρει ε, πότε και αν θα υπάρξει νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ορίσατε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε πρώτον και δεύτερον σας ευχαριστούμε διότι καταφέρατε να έρθετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μήνυ Υπουργικής Συνόδου στη Σανγκάη. Ε, τη μία στιγμή ήσασταν εκεί, την άλλη στιγμή είστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Άρα μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της μήνυ Υπουργικής Συνόδου στη Σανγκάη και κυρίως μπορείτε να μας ενημερώσετε και για την υπουργική διάσκεψη τον Ιούνιο του 20 στο Καζακστάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ακόμα εδώ. Νόμιζα ότι θα είναι τελευταία η προηγούμενη φορά, μπορεί να είναι αυτή. Αν όχι, θα με ευτυχής να ξαναέρθω. Πράγματι, μόλις ε, επέστρεψα από την ε, Σανγκάη, υπήρχε αυτή η μην υπουργική διάσκεψη για να γίνει ένας απολογισμός της κατάστασης στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που μάλλον θα πάψει να υπάρχει, θα υποστεί σημαντικές απώλειες σε κάμια δύο εβδομάδες και θέλαμε να δούμε τι μπορεί να γίνει ε, για την υπουργική διάσκεψη του Ιουνίου στο Καζακστάν. Το πιο ε, σημαντικό ζήτημα, όπως σας είπα, είναι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που δεν θα μπορεί πλέον να επιλαμβάνεται νέων προσφυγών μετά τις 10 Δεκεμβρίου, διότι ε, δεν θα ε, μπορέσει να εγκριθεί νέα, δεν θα μπορέσουν να εγκριθούν νέα μέλη, εκ η θητεία των τριών τελευταίων ή παρνούνται να ορίσουν ε, κάποιον και έχουμε τον Αμερικανό που επειδή μπορεί να μην παραμείνει σε αυτό το όργανο δεν μπορεί να εξετάσει τις εκκρεμούσες υποθέσεις και μπορεί η επίλυση να γίνεται με τα πάνελ, κάτι που όπως ξέρετε δεν είναι ευκταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο και όλα τα κράτη-μέλη είναι ενωμένοι στην προσέγγιση τους. Στηρίζουμε τη διαδικασία που δρομολογήθηκε ε, από τον ε, πρέσβη Γόκερ της Νέας Λανδίας για την ε, ε, λύση του αδιεξόδου. Η πρέσβηση ε, πρότεινε κάποιες ε, δυνατότητες για τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και για την πλήρωση των θέσεων που χειρεύουν και παρουσιάστηκε στην πρόσφατη γενική, συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων το Δεκέμβριο. Το... είπα όμως δεν ήθελα να συμμετέχουν, συμμετέχουν άσκησαν κριτική αλλά οι άλλοι 163 ε, από τον ΠΟΕ μπορούν να δεχθούν αυτή την πρόταση. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις, υπάρχει λοιπόν υποστήριξη. Δεν υπήρξαν, κοινές, ε, δεν υπήρξαν κοινά συμπεράσματα. Ελπίζουμε ότι οι ΙΠΑ θα μπορέσουν να υποστηρίξουν στο τέλος. Δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη βέβαια, δυστυχώς. Όπως γνωρίζετε, βρήκαμε μια ενδιάμεση λύση για να εκπροσωπήσουμε τα δικά μας δικαιώματα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ, διάμεση, ε, διμερής αν θέλετε προσέγγιση με ανεξάρτητους δικαστές, ε, παλαιούς δικαστές του ΠΟΕ και με τη βοήθεια της γραμματείας για να έχουμε έτσι μια αμοιβαία ε, διευθέτηση διακανονισμό μέχρι να ξανακαταστεί επιχειρησιακό το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο. Δεν είναι ιδέα τη λύση, αλλά η Νορβηγία και ο Καναδά συμφώνησαν, έχουμε πολλά συμφωνία και απευθυνόμαστε και σε άλλες χώρες ε, και ιδίως αυτές με τις οποίες ε, έχουμε διαμάχη και αντιπαράθεση. Στόχος είναι να έχουμε πλείονα μέρη, αλλά προς το παρόν Έχουμε συνομιλίες, αλλά η συμφωνία ε, είναι μόνο με αυτές που σας ανέφερα, τις δύο. Ως βλέπουμε την 12η ε, Υπουργική Διάσκεψη, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Πάντως θα είναι ένα μετέχνη για να δούμε κατά πόσο ο ΠΟΕ θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει τα αποτελέσματα που πρέπει και να κάνει και σοβαρές προσπάθειες για να ε, συνεχίσει δεν ξέρω αν είναι η στιγμή να καταθέσουμε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό πακέτο, έστω να συμφωνήσουμε σε κάποια σημεία για να ξεκινήσει μια μεταρρύθμιση. Αυτό θα ήταν καλό. Τρει είναι οι τομεί όπου θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τη βιωσιμότητα, αν θέλετε, του ΠΟΕ, ως επίκεντρο του πολυμερού συστήματος εμπορίου. Καταρχά, όπω γνωρίζετε, ε, κάνουμε προσπάθειες κατάρτισης κανόνων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου υπηρεσιών αλίας και τα λοιπά ή ε, επιδοτήσεις στον τομέα της αλίας. Υποτίθεται ότι θα είχαμε κλείσει το θέμα αυτό μέχρι τα τέλη του έτους. Δεν θα συμβεί αυτό. Όμως ε, διαπραγματευόμαστε, είναι σε εξέλιξη όλες αυτές οι συνομιλίες, αλλά δεν ε, έχει οριστεί ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας ακόμη. Ελπίζουμε αυτό να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ήταν άκρος λυπηρό να μην καταλήξουμε σε συμφωνία. Γιατί αν συμφωνήσουμε θα στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι το εμπόριο, η βιώσιμη ανάπτυξη συμβαδίζουν, πάνε χέρι-χέρι. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται, είναι όμως δύσκολες. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ε, δυνατότητα να έχουμε συμφωνήσει. Το Μάιο τώρα φέτο 59 μέλη του ΠΟΕ ενέκριναν μια δήλωση για έναν κανονισμό για τις υπηρεσίες ε, στο πιστόσα του το Παρίσι. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ε, έντονες επαφές ε, και την προηγούμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα θα πετύχει εδώ η διαπραγμάτευση, αν προχωρήσει όπως προχωρά, θετικά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο γίνονται διαπραγματεύσεις, προχωρούν δεν ξέρω αν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, αλλά θα μπορούμε νομίζω να έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο. 92 χώρε έχουν πει ότι θέλουν να συμπεριληφθούν στι διαπραγματεύσει για τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Το ανακοίνωσε χθε η Κινέζικη Προεδρία. Και εδώ έχουμε πρόοδο. Θα δούμε πού βρισκόμαστε τον Ιούνιο. Και ίσω ε, η απαγόρευση, το μορατόριο ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να ανανεωθεί τον Ιούνιο. Ε, πολλοί υπουργοί χθε είπαν ότι και στον τομέα των κοινών πρέπει να κάνουμε πρόοδο, αλλά λίγα συγκεκριμένα ζητήματα ετέθησαν. Θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι προτάσεις θα κατατεθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με άλλους κατέθεσε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διαδικαστικών ε, πτυχών, για τις κοινοποιήσεις, προτάσεις ε, κτλ. Και τρίτον, κάνουμε προσπάθειες για να έχουμε δικούς κανόνες παιχνίδι στο μέλλον, δηλαδή ε, επιδοτήσεις, ε, μεταφά τεχνογνωσίας, με υπαϊπονία εργαζόμαστε και μεταρρύθμιση ειδική δεκτικής μεταχείρισης, πολύ ακαθόδης θέμα. Τα δύο τρίτα όμως τώρα των κρατών μελών αποκλείονται, ξερούνται από τους κανόνες δεν υπακούν στις ίδιες ε, προποθέσει και διαδικασίες διαφάνειας, κοινοποίηση, Αυτό δεν θέλουμε να ισχύει. Ε, από την Ορβηγία ο Υπουργό κάνει κάποιες προσπάθειες και θα προσπαθήσουμε να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ίσως αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε καταγράψει μέχρι τον Ιούνιο και ίσως να έχουμε ολοκληρώσει με φορισμένων από αυτόν. Θα δούμε αλλά δεν νομίζω να πετύχουμε τις δραστικές μεταρρυθμίσεις του ΠΟΕ άμεσα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει για να παραμείνει στο επίκεντρο. Υπάρχει συμφωνία σχετικά, πολύ λίγες όμως συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες προτάσεις για ε, να μην δουλεύουν σε πολυμερές, αλλά σε πλειομερές ε, επίπεδο. Δεν βλέπουμε όμως αντίστοιχη αίσθηση κατεπήγοντος για το θέμα αυτό και από άλλους. Ε, άρα αυτό είναι ένα θέμα θα το δούμε και του χρόνου ε, για να δούμε τι μπορεί να είναι ρεαλιστικό. Αν θα στείλουμε στο Πακιστάν, ε, μάλλον στον Παγκλαντές, ε, την αντιπροσωπεία μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε εσείς κάτι, μάλλον αν θέλετε να πω κάτι για τη ΣΥΠΑ και τους δασμούς. Με τα χαράς, λέει ο πρόεδρος. Ε, με τα χαράς, δεν ξέρω, αλλά... πολύ χρόνο δαπανίσαμε για να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο για τα εμπορικά θέματα με τη ΣΥΠΑ. Έχουμε διαφωνίες όμως είναι παρόλα αυτά ο πιο σημαντικός εμπορικός επενδυτικός μας εταίρος. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις εμπορικές εντάσεις και να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο. Ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Ιούλιο πήγε στην Ουάσιγκτον και στάνε στον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχουμε πολλά σκέλη, πολλούς άξονες. Έχουμε την έκθεση προόδου που δημοσιεύσαμε πριν από δύο-τρει μήνες ε, και εκεί λέμε ότι θέλουμε για τη συμμόρφωση ε, και για τα πρότυπα, νέες τεχνολογίες όπως η ρομποτική, η, η εκτύπωση. Θέλουμε πρόοδο και έχουμε καταθέσει προτάσεις, χωρίς να υπάρχει ακόμη συμφωνία. Προοδεύουμε όμως. Δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια πιο περιορισμένη υπορική συμφωνία, πιο περιορισμένη για τα βιομηχανικά αγαθά και την αλία, αυτή είναι η εντολή που μα δόθηκε, πιο μικρέ κλιμάκα, περιορισμένη συμφωνία. Εμεί είμαστε έτοιμοι, αλλά οι Αμερικάνοι δεν έχουν κάνει κάποιο βήμα από την πλευρά του μέχρι στιγμή. Έχουμε επίση εργαστεί ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα πιστοποίηση μόρφωση και αξιολόγηση μόρφωση. Κάποια πρόοδο υπάρχει, δεν έχουμε όμω φτάσει ικανοποιητικό επίπεδο και πολύ πρόοδο θα έλεγα έχουμε επιτελέσει στην μεταρρύθμιση του ίδιου του εμπορικού συστήματο. Ξέρετε ε, ότι υπάρχουν κάποιες κριτικές από τις ΗΠΑ κατά της Κίνας. Συμφωνούμε, αλλά δεν συμφωνούμε με τη μέθοδο. Θέλουμε πολυμερή προσέγγιση, θέλουμε κανόνες για την εξαναγκαστική μεταφορά τεχνογνωσίας ή ε, τις βιομηχανικές επιδοτήσεις. Ε, οι εργασίες μας είναι εντατικέ, ανταλλάσσουμε έγγραφα, δεν έχουμε ακόμη κάποια έτσι, ικανοποιητική εξέλιξη, αλλά ελπίζουμε σύντομα. Επίσης, όπως γνωρίζετε, είχαμε την διαμάχη Airbus Boeing με τη ΣΥΠΑ. Από τις 18 Οκτωβρίου επίσης επιβάλλουν δασμούς σε κάποια προϊόντα ε, και πριν από δύο εβδομάδες το συζητήσαμε στην Ολομέλη αυτό. Το συζήτησα με τους πρέσβεις και είπα ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί λύση γιατί θα μπορέσουμε, ε, θα έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε και εμείς δασμούς για το χρόνο αυτό. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση στο μεταξύ. Την έννοια των διαπραγματεύσεων δεν την έχουν απορρίψει, αλλά δεν βιάζονται. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει αυτή η μακροχρόνια διαμάχη, 16-17 έτη, να ε, τυλίξουμε κάποια στιγμή γιατί έχουν ε, βγάλει πολλά λεφτά δικηγόροι από αυτή την υπόθεση όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε και νέους ε, παίκτες στην αγορά της αεροναυπηγικής. Επίσης έχουμε δικαιολόγητα μέτρα κατά της εισαγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Είχαμε μια εξάμεινη παράταση, αναβολή ε, εμείς έχουμε πει ότι είμαστε εταίροι και θέμα της ασφαλείας. Οι εξαγωγές ε, οχημάτων ή ανταλλακτικών εξαρτημάτων οχημάτων δεν απειλεί την ε, εθνική ασφάλεια των ήπα, Γιατί αυτοί με αυτό το άρθρο το 232 για την εθνική ασφάλεια δικαιολογούν τα μέτρα που θέλουν να λάβουν. Έχουμε τατικές συζητήσεις και ξέρω ότι και ευρωβουλευτέ το ίδιο μήνυμα έχουν επαναλάβει ότι δεν θα ήταν καλό για εμά, αλλά ούτε και για τη ΣΥΠΑ διότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί πολλούς και στη ΣΥΠΑ, που σημαίνει ότι και αυτοί θα πληγούν. Είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε τους δασμούς ε, στα οχήματα, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας για τα βιομηχανικά αγαθά και ότι μπορούμε να συστήσουμε και τα πρότυπα για να έχουμε την ευκαιρία να προβούμε σε μια αριθμιστική σύγκληση, να είναι πιο συμβατά τα πρότυπα. Αυτό είναι θετικό και για τις δύο πλευρές. Δεν γνωρίζουμε τι θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα. Ε, διάφορα δημοσιεύματα αντιφατικά μεταξύ τους ε, κυκλοφορούν. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που από ό,τι φαίνεται στηρίζουν ε, την ιδέα δασμών για το τομέα των αυτοκινήτων. Θα συνεχίσουμε τις επαφές μας μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και έχουμε πει επίσης ξεκάθαρα ότι εθελοντικές εξαγωγές ή εθελοντικές διατάξεις και συμφωνίες δεν είναι συμβατές με τον ΠΟΕ. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε αποφασιστικοί, κατηγορηματικοί και αν υπάρξουν νέοι εμπορικοί περιορισμοί θα ε, ληφθούν μέτρα επανεξισορρόπησης που σίγουρα θα πλήξουν την θετική ατζέντα, το θετικό θεματολόγιο. Ε, κάτι θετικό για να κλείσω λύσαμε τις διαφορές μας με το βόλιο κρέας. Ε, νομίζω το συστήσατε κι εσείς. Ε, ελπίζω να ψηφίσει ε, θετικά το Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Παλαιά και αυτή, έχει χρονίσει. Καλό θα ήταν να κλείσει το θέμα αυτό. Δεν θα επηρεάσει τις ποσοστώσεις κρέατος που εισάγεται στις ευρωπαϊκές αγορές. Νομίζω ότι το θετικό είναι ότι ήταν ενωμένα τα κρατημέλη, η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρότι είναι δύσκολη κατάσταση. Μία ευρωπαϊκή φωνή ακουγόταν, το ίδιο μήνυμα λίγο πολύ, ίσως με διαφορετικό τρόπο, αλλά το ίδιο μήνυμα και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον να πορευόμαστε. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, να είμαστε αυστηροί, σκληροί, ενωμένοι και βασόμαστε την Κομισιόν γι' αυτό. Ιδίως για τα αυτοκίνητα μέχρι τελευταία στιγμή πρέπει να υπερασπίσει τα συμφέροντά μας και να προβάλλει τα δικά μας επιχειρήματα, τις δικές μας θέσεις. Δύσκολη επίσης και σημαντική παρόλα αυτά η μάχη για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ που θα κυριαρχήσει πιστεύω στα εμπορικά συστήματα του χρόνου και η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντική. Σταματώ εδώ και είμαι διατεθειμένη και έτοιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σεσίλια. Αρκετά έχουν ζητήσει το λόγο. Ο Κρίστοφ. Κρίστοφ Χάνσεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πέρντ. Ευχαριστούμε Σεσίλια που βρήκε το χρόνο και ήρθες και πάλι πίσω στις Βρυξέλλες για να είσαι κοντά μας. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που είχα κατά το παρελθόν την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου, κυρίως ε, για το πολύ ενδιαφέρον θέμα από την τελευταία ε, θητεία ε, συμφωνία με την Ιαπωνία. Ο κύριος Περέιρα ήταν ο εισηγητής, ο κύριος Σίλβα Περέιρα και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια πολύ σημαντική εξέλιξη και χαίρομαι που βρίσκει σήμερα εδώ. Νομίζω αυτή είναι και η τελευταία σου ε, συνάντηση με την Επιτροπή μας, με την ιδιότητά σου της Επιτρόπου Εμπορίου. Μας αφήνεις όμως σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις ε, μπροστά μας, ε, τα, μαζεύονται τα σύννεφα, τα σκοτεινά σύννεφα στον ορίζοντα. Ε, και νομίζω ότι θα υπάρξουν δυσάρες εξελίξεις για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που εκκρεμούν με τις ΗΠΑ. Η υπόθεση Airbus, η απόφαση ε, σε επίπεδο ΠΟΕ ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση γιατί ε, δώσαμε παράνομες επιδοτήσεις ε, στου κατασκευαστές, αλλά απ' την άλλη και οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν ακριβώ το ίδιο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην ε, πυροβολεί ο κάθε ένας από εμά τον άλλον στο πόδι του, γιατί υπάρχουν ε, και οι που καραδοκούν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα τα χάσουμε τελικά όλα αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να βρούμε, να αναζητήσουμε κάποια διεθνώς αποδεικτή λύση για τις ε, επιδοτήσεις ε, στους ε, κατασκευαστές αεροσκαφών. Κατά τα άλλα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση. Αναφερθήκατε στις ε, ποσοστώσεις, στις δασμολογικές ποσοστώσεις για το βόλιο κρέας. Και αυτό από πλευρά μας είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα και ένα μήνυμα ότι παραμένουμε πιστοί στις υποχρώσεις μας ε, στον ΠΟΕ. Ελπίζω αυτό να περάσει στις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί νομίζω ότι εκείνοι ε, καταφεύγουν σε αυτές τις αποφάσεις, αλλά εν πάση θα πρέπει να υπάρχει μία συνέπεια. Νομίζω ότι ο ΠΟΕ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ε, διεθνούς εμπορίου. Ολοκληρώνω, γιατί βλέπω και το σφυράκι του Μπέρντ να με ε, στοχεύει. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ψήφισμα ότι είμαστε υπέρ της λειτουργίας ε, του ΠΟΕ και επιθυμούμε να υπάρχει ένα ε, δευτερογενές δικαιοδοτικό όργανο το οποίο να ρυθμίζει και να παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, γιατί υπάρχει και άλλη μια συνάντηση της Επιτροπής 25 και εκεί ε, μπορούμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα που να εγκριθεί κιόλα ε, κατά τη διάρκεια ε, τη Συνόδου. Και ίσω οι συνάδελφοι μπορούν να μου πούνε αν συμφωνούν με αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, δώσουμε ένα μήνυμα πριν από τις 10 Δεκεμβρίου ότι πραγματικά επιθυμούμε να υπάρχει ένας επικοδομητικός διάλογος για τις ε, μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθεί αυτό το κόσμημα ε, που υφίσταται και που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μαρή Βεντρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Καλώς ήλθατε από τη Σανγκάη. Προλίγου Ήμουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων από τη Βρετάνη και ένας από αυτούς μου είπε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να μιλήσει για τα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, δική μας περιφέρεια και δεν βλέπει καθόλου το θετικό αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του. Εγώ λοιπόν ε, έβγαλα μεγαλεπίβολη ομιλία για τις διεθνείς συμφωνίες για το πόσο μπορεί να ωφεληθεί η Βρετάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τον έπεισα όμως και βλέπετε ε, τους λαϊκιστές να ανεβαίνουν παντού στην Ευρώπη. Ως αιρετοί με καθολική ψηφοφορία έχουμε διπλή ευθύνη και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια και εμείς. Έχουμε την ομάδα παρακολούθησης και εποπτείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και νομίζω ότι μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα και στον ΠΟΕ. Ποιο είναι το όραμά σας, ποιες είναι οι συμβουλές σας. Ίσως είναι και η τελευταία φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας με αυτή σας την ιδιότητα. Πώς θα υπερασπιστούμε ένα εμπόριο δίκαιο ισορροπημένο, που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Θα μπορούσα να σας θέσω διάφορα άλλα ερωτήματα τεχνικά, όμως έχουμε και πολιτική ευθύνη, ξέρετε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να υπερασπιζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το όραμά της. Έχει αληθινό όραμα η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σίλβα Περέιρα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δράξω αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ την Επιτροπό μας, να τη συγχαρώ για την εξαιρετική της επίδοση ως Επίτροπος ε, βοήθησε στο να έχουμε μια φιλόδοξη, ε, φιλόδοξα, να αντιμετωπίσουμε φιλόδοξα θέματα ως Επιτροπή Εμπορίου. Ε, μην ξεχνάμε ότι ήταν, μενόταν ένα εμπορικός πόλεμος σε πάρα πολλά θέματα. Είχαμε βέβαια την συμφωνία με τον Καναδά, αλλά κυρίως τη συμφωνία με την Ιαπωνία, όπου εγώ ήμουν εισηγητής. Και νομίζω ότι είναι η σημαντικότερη εμπορική συμφωνία που συνήφθη ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα έρχεστε εδώ σήμερα για να μας μιλήσετε για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Ε, για άλλη μια φορά, είσαστε στην ε, σωστή πλευρά των εξελίξεων. Ε, αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, της πολυμέρειας και του εμπορίου, του ευνομούμενου εμπορίου, σωστή είναι αυτή η κατεύθυνση. Όσον αφορά στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μία βέβαια πρέπει να είμαστε σταθεροί, γιατί πράγματι πρέπει να είμαστε σταθεροί, όμως οφείλουμε να αναζητήσουμε και θετικά θέματα. Τώρα λοιπόν που σημειώνεται πρόοδο σε αυτά τα θετικά ε, θέματα, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στην πορεία μας. Τελειώνοντας να πω ότι ε, δεν ξέρω, βλέπετε εσείς να υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα στο, στην καθυστέρηση που προκύπτει με τον ε, διορισμό της Νέας Επιτροπής, εκτός από το ότι έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε περισσότερο. Κυρία Επίτροπε, θέλω και εγώ να σας ε, συγχαρώ ε, για την ε, πολύ καλή θητεία σας. Πολλές συμφωνίες συνήφθησαν και πάρα πολλές έπονται Πράγματι υπήρχε διαφάνεια, υπήρχαν συζητήσεις με τα κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά και σας ευχαριστώ και για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ κυρίως για τις προσπάθειές σας να σώσετε τον ΠΟΕ. Ε, νομίζω αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλους μας. Και ήταν πολύ καλό αυτό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποίοι ε, εργάστηκε για έναν εναλλακτικό μηχανισμό για το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο. Σας συγχαίρουμε για τις προσπάθειές σας να εξυγχρονίσετε τον ΠΟΕ. Έχω μία ερώτηση που αφορά στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, περισσότερες πληροφορίες. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Απομακρύνονται ουσιαστικά από τη μονομέρεια και πηγαίνουν προς την πολυμέρεια ή προς τον απομονωτισμό. Ε, τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν ε, πιστεύετε όπως είπε και η πρόεδρος της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, αν πιστεύετε κι εσείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο ε, για να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να σας πω ότι εμείς ε, θα στηρίξουμε το ψήφισμα. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο που μόλις προσγειώθηκε, έτρεξε εδώ, σε εμά. Ε, πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι κανοποιημένος που λέτε ότι ε, θα προσπαθήσετε να βρείτε μια εναλλακτική λύση για να λύσετε αυτό το πρόβλημα των ε, δευτεροβάθμιων, ε, του δευτεροβάθμιου διοικητικού δικαιοδοτικού οργάνου. Πάντως το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Άρα δηλαδή, επειδή ίσως υπάρχει άλλη μια ευκαιρία για να συζητήσουμε. Μήπως θα πρέπει τα θέματα να τα τοποθετήσουμε διαφορετικά. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Ε, συνάντηση κορυφή στη Νέα Υόρκη. Σε πολλές ε, περιπτώσεις λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εργασίας μας. Και αυτό ε, συμπεριλαμβάνει και τον ΠΟΕ. Από την εμπειρία σας λοιπόν των τελευταίων 5 ετών. Πού ακριβώς πιστεύετε ότι μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε διαφορετικά θέματα. Γιατί αν ένα θέμα δεν καρποφορεί πρέπει να το αλλάξουμε και να επιλέξουμε διαφορετικά θέματα. Εσείς λοιπόν τι έχετε να ε, συστήσετε, τι συστήνετε ε, με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα στον ΠΟΕ. Τώρα ο κύριος Κασπάρη. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, αγαστή συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Αν δούμε λιγάκι πού ακριβώς βρισκόταν η εμπορική πολιτική και ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα ε, δέκα χρόνια Μάντελσον, Άρσον και Ντεκούχτ. πράγματι είχατε ε, πολλέ δυσκολίε να αντιμετωπίσετε. Κατορθώσατε όμως να συνάψετε εμπορική συμφωνία και κυρίως εδώ να ε, εμπνεύσετε ε, με εμπιστοσύνη. Ε, αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Όσον αφορά στα θέματα που θίξατε, συγκεκριμένα τώρα. Ε, σε, αυτή, σε αυτές τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΠΟΕ. Ε, να σας πω ειλικρινά ότι μετά την τελική διακήρυξη που δημοσιεύτηκε νιώθω απογοητευμένος. Ε, βεβαίως γιατί δεν συμμετέχουν οι Αμερικανοί όπως θα έπρεπε. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε ε, δημιουργήσει μια γέφυρα όπου κατ' ουσίαν θα τους αναγκάζουμε να δεσμευτούν για πολυμέρεια και πολυμερείς σχέσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Χάνσεν είναι πολύ καλή πρόταση να τοποθετηθούμε δηλαδή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως σας ρωτώ, εσάς, πιστεύετε ότι υπάρχει ίσως κάτι όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει κάτι για να ασκηθεί ε, μεγαλύτερη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να δεσμευτούν έναντι του ΠΟΕ, κυρίως έχοντας ε, κατά νου τις μεταρρυθμίσεις που επίκυνται. Ε, πιστεύετε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα έτσι ώστε να ε, ξεμπλοκαριστεί το όλο θέμα των ε, διτητικών δικαστηρίων. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτησή σας ε, για το πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ, κυρία Επιτροπέ, που ήρθατε εδώ να μας δείτε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την κληρονομιά και η κληρονομιά της Επιτροπής Γιούνκερ θα είναι αμφίσιμη. Είναι δύσκολο να έχουμε ξεκάθαρη αξιολόγηση αυτής της κληρονομιάς. Το εμπόριο όμως ήταν ένας από τους τομείς που η Επιτροπή Γιούνκερ έφερε εξαιρετικά αποτελέσματα, άρα και εσείς και η δική μας Επιτροπή ε, συνεργάστηκε μαζί σας με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συμφωνώ με τον Ντανιέλ Κάσπαρη και το λέω για τους νέους συναδέλφους. Δεν θα μάθουν ποτέ πώς ήταν η κατάσταση πριν από 6-7 χρόνια. Μετά από μια περίοδο διαλόγου εξαιρετικά σημαντική, Είχαμε διάφορες ιδέες και τις συζητήσαμε μαζί σας, Επίτροπε για τη διεύρυνση του πεδίου ερμοδιοτήτων της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στα χωράφια της παρακολούθησης και της εποπτείας των συμφωνιών που συνάπτουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή τους. Αυτό είναι το μεγάλο πεδίο, το επόμενο μεγάλο βήμα. Δεν έχω ερωτήσει να σας θέσω, θέλω να σας συγχαρώ θερμά κύριε Επίτροπε και να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ κυρία Ροντρίγκε Πιέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι η συντονίστρια της ομάδας μας, η Κάθλιν Βαν Μπρέμτε, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Και νομίζω ότι η γραμματεία το ήξερε αυτό. Επομένως, σας συγχαίρω εξ ονόματος της κυρίας Μπρέμτε, αλλά και ε, εγώ η ίδια. Θέλω να σας ευχαριστώ για τη στάση που είχατε και εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο και τη στάση που είχατε με τις τρίτες χώρες. Γνωρίζουμε τη δραστηριότητα σα υπερασπίζεστε πάντοτε τι εμπορικέ συμφωνίε. Δυσκολεύεστε βεβαίω να... θέλετε πάντοτε και έχετε πολύ αγωνιστεί να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στι εμπορικέ συμφωνίε. Π.χ. Ε, στη συμφωνία με τον Μπαγκλαντέ, ε, βάλατε την κατάργηση των ε, αγαθών διτής χρήση, την κατάργηση των προϊόντων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή εργαλείων βασανιστήριων και Πιστεύω ότι πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με το έργο που έχετε υλοποιήσει ε, γενικά και όλοι γνωρίζουμε πόσο προσιλωμένοι ήσασταν σε αυτά τα θέματα. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί. Πιστεύετε ότι αν υπάρχει συμφωνία με την Κίνα θα αλλάξει η στάση των ΗΠΑ. Σε ποιο βαθμό ασκείται αυτή η πίεση στον ΠΟΕ που τον καθιστά παραλυμένο τελικά οργανισμό που να μην μπορεί να δράσει. Μπορεί όλο αυτό να είναι ένα έξτρα στοιχείο άσκησης πίεσης στην Κίνα. Μπορεί τελικά να καταλήξουν σε συμφωνία ΙΠΑ και Κίνα και να αρχίσει να υπάρχει μια κατάσταση εμπιστοσύνης η οποία ε, μπορεί να υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες για να υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, με όλες αυτές τις αβεβαιότητες και αμφιβολίες ε, για τη μεταρρύθμιση στην Υπουργική Διάσκεψη πιστεύετε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε διαφορετική κατάσταση όπου να μην υπάρξει τελική διακήρυξη όπου όσο έγινε και στον Buenos Άιρε θα υπάρχει σχέδιο Β στο Buenos Aires δεν υπήρξε κοινή διακήρυξη, αλλά υπήρχε διακήρυξη για θέματα του φύλου, την οποία προσυπέραψαν διάφορες χώρες. Έχουμε ένα σχέδιο Β. Αν δεν υπάρξει κοινή δήλωση, να υπάρξει κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές, έτσι ώστε να, δώσουμε το, να εκφράσουμε το μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι συζητούμε και είμαστε ικανοί να καταλήξουμε κάπου. Και τρίτον, για τα δασμολογικά θέματα. Μπορεί να υπάρξουν ενισχύσεις στο γεωργικό τομέα, ο οποίος πλήττεται από μείωση δασμών για λόγους που για τους οποίους δεν ευθύνεται. Θεωρείτε πραγματικά ότι αυτό το κοινοβούλιο, πέρα από το ψήφισμα, το οποίο είναι πολύ καλή πρωτοβουλία βεβαίως, και θα το υποβάλουμε στην επόμενη Ολομέλεια. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω αυτό το Κοινοβούλιο για να ενισχύσει και να βοηθήσει ε, ε, στη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Για το Renew παρακαλώ. Καρίν Κάρλσμπουργκ. Σας ευχαριστώ. Θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να σας πω το εξής. Ευχαριστώ Σεσίλια και ευχαριστώ εσένα και την ομάδα σου για όλα όσα κάνατε. Ήσουν επίτροπος και είσαι επικεφαλής αρμόδιος για θέματα εμπορίου και εγώ εκπροσωπώ το σύνολο της πολιτικής μας ομάδας. Πιστεύουμε ότι είσαι καταπληκτική. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για σένα, για όλα αυτά τα οποία έκανες, για όλες αυτές τις προσπάθειες που κατέβαλες, για ένα ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο παγκοσμίω. Νομίζω ότι εσύ άλλαξε την εμπορική πολιτική παγκοσμίω και μάλιστα πολύ. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι, διότι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για κεφάλαια, κεφάλαια αηφορίας. Ε, στις εμπορικές συμφωνίες και να απαντούμε αυτό στους ανθρώπους που μας λένε ότι η κλιματική αλλαγή και η ανισότητα των φύλων οφείλονται εν μέρη στο εμπόριο. Και εμείς έχουμε απάντηση να δώσουμε. Επιτέλους, χάρη σε σένα. Υπήρξε σύνδεση με το, μεταξύ εμπορίου και ε, κλιματικής αλλαγής και λοιπόν προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Σε ξέρω, σε γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι ε, είσαι αταλάντευτα προσιλωμένη στην ανοιχτή κοινωνία, στις αξίες που έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φίλων. Θα κλείσω κάπου εδώ ζητώντας σου να μας δώσεις κάποιες συμβουλές. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εμπορική ε, ε, πολιτική όταν προβάλλουμε το επιχείρημα για περισσότερο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και για περισσότερες δημοκρατικές εξελίξεις στον πλανήτη μας, θετικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα και για χώρες που δεν είναι στη θέση την οποία, στην οποία θα θέλαμε να βρίσκονται σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Χιούμπνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω κι εγώ πολλά να πω. Προσυπογράφω πλήρως. Ε, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες για όλα όσα υπόθηκαν για σένα, Σεσίλια. Λυπάμαι για τον Φιλ Χόγκαν, γιατί θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για αυτό να καλύψει το κενό που αφήνεις με την αναχώρησή σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Έχω δύο δύσκολα ερωτήματα να σου θέσω ωστόσο. Η κατάσταση το Δεκέμβριο που θα έχουμε στον ΠΟΕ, ποια είναι. Ε, κάτι δεν γνωρίζω, κάτι αγνοώ, κάτι δεν έχω καταλάβει. Μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο και να οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση τη στιγμή κατά την οποία θα έχουμε τα στοιχεία για την Boeing. Υπάρχουν, υπάρχει κάποια διαδικασία διαιτησίας ή είναι διαφορετικό το όργανο αυτό. Επίσης αναφερθήκατε, αναφέρθηκε στον Καναδά και στην Νορβηγία και στις προσπάθειες να καλυφθεί αυτό το κενό όπου δεν έχουμε αρμόδιο όργανο με ενδιάμεση φόρμουλα και είπατε ότι εξετάζετε και άλλους εταίρους και τις συμφωνίες με άλλους εταίρους, μήπως μπορείτε να εμπνευστείτε από εκεί. Όμως δεν υιοθετούν και άλλα μέλη του ΠΟΕ αυτή την προσέγγιση. Σκέφτονται να φτιάξουν κάτι αντίστοιχο με τους δικούς τους εταίρους, όχι με εμά. Είναι επινόηση μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό και πρωτοβουλία μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιουτικόφερ παρακαλώ τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για τη δουλειά σας. Συμφωνώ απολύτως με ε, τε, τους επένους, τους πράγματι δικαιολογημένους που σας επιφύλαξαν οι προλαλήσαντες. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, αυτή είναι η πρότιμη παρατήρησή μου. Είπατε ότι πρέπει να ε, ασκήσουμε πίεση στη ΣΥΠΑ. Τέτοιου είδους διατυπώσεις δεν βοηθούν κατά την άποψή μου. Στις Πολιτείες είναι διαφορετικοί οι παράγοντες και δεν είδα κανέναν να ασκεί πίεση επιτυχώς στον πρόεδρο Τραμπ μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο μόνος άνθρωπος που πράγματι κατάφερε να επιτύχει μια καλή συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ ήταν ο πρόεδρος Γιούνκερ και δεν το κατάφερε ασκώντας πίεση στον πρόεδρο Τραμπ και αυτό το έχει περιγράψει σε συνέντευξή του. Προτείνω να αντλήσουμε διδάγματα από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Ε, υπάρχουν όμως και άλλοι παίκτες και άλλοι παράγοντες της ΣΥΠΑ και δεν είναι η σωστή προσέγγιση να τους ασκούμε πίεση, αλλά η σωστή προσέγγιση είναι να βρίσκουμε κοινό έδαφος με αυτούς τους ανθρώπους. Μίλησα με συνομιλητές την περασμένη εβδομάδα στη Ουάσιγκτον και πολλοί μου είπαν το εξής. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι κατά των δασμών. Οι οργανώσει των επιμελητηρίων είναι κατά και οι διοικητέ κυβερνήτε των πολιτιών είναι κατά και διάφοροι ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο είναι κατά. Άρα δεν είναι ο σκοπός, δεν είναι χρήσιμο να ασκήσουμε πίεση, αλλά να συνάψουμε συμμαχίες για να αναδείξουμε τις απόψεις μας. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση μας τώρα για την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και πιο συγκεκριμένα για το σώμα που εκδικάζει τις προσφυγές. Συμφωνώ να μπει αυτό στην ημερήσια διάταξη όπως προτάθηκε, συμφωνώ απολύτως. Δεν θα είχε νόημα να μπούμε σε λεπτομέρειες, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, ένα πολιτικό σινιάλο ότι είναι ε, ζήτημα εξέχουσας σημασίας, επιμένουμε σε αυτό, θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτό το όργανο και συνάμα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τη ΣΥΠΑ για να επέλθουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η προσέγγιση μου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Δίνω το λόγο αμέσως στη Σεσίλια. Σα ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για μένα ήταν πολύ μεγάλη απόλαυση να μπορώ να συνεργάζομαι μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι εμεί και και εσείς πετύχαμε πολλά καλά πράγματα μαζί. Δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά άποψή μου είναι ότι είναι καλό να βγάλετε ψήφισμα για αυτό το σώμα εκδίκασης προσφυγών στο πλαίσιο του ΠΟΕ ε, και είμαι ε, ότι θέλουμε να επιζήσει αυτό και μπορούμε να συζητήσουμε και μεταρρυθμίσεις. Και πολλά μένει να συζητηθούν στην Υπουργική Διάσκεψη του Ιουνίου. Όμως μπορείτε να καθυστερήσετε ένα τέτοιο αντίστοιχο ψήφισμα για την Άνοιξη, για να ε, υπάρξουν και προτάσεις και να τις εμπεριλάβετε. Το πιο τρέχον και επίγον αυτή τη στιγμή είναι αυτό το σώμα ε, εξέτασης των προσφυγών. Κύριε Μπουρζουά, για τα ερωτήματά σας, δεν νομίζω ότι η πολυμερής προσέγγιση είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις στις ΗΠΑ, σωστά το λέει ο κύριος Beauty Coffer. Η τρέχουσα κυβέρνηση στη ΣΥΠΑ ε, θέλει τις διμερείς συμφωνίες, δεν συμφωνεί με την πολυμερή προσέγγιση και άρα η πολυμερή προσέγγιση περιορίζει τις δυνατότητες και το περιθώριο ελιγμών για την κυβέρνηση, θεωρούν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, ο ΠΟΕ είναι καλός ε, για τις ΗΠΑ, έχουν κερδίσει πολλές υποθέσεις στο ΠΟΕ, στα διάφορα δικαστήρια του ΠΟΕ και έχουν διάφορες ασκήσεις ε, πειθάρχησης που έχουν επιβάλει για τη θέσπιση κοινών κανόνων, για την κατάργηση δασμών. Όλα αυτά τα έχουν κάνει μέσα στο ΠΟΕ, έχουν γίνει στο παρελθόν εντός των ΠΟΕ και πρέπει αυτό το μήνυμα να το στέλνουμε ξανά και ξανά. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συνεχίσουν τις επαφές τους με το Κογκρέσο στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν πάρα πολλά μέλη του Κογκρέσου, πάρα πολλοί γερουσιαστές που είναι πεπισμένοι ευρωατλαντιστές, που πραγματικά πιστεύουν ότι η φιλία, οι στέρεες σχέσεις, οι στενές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΕΕ είναι κάτι το σημαντικό, κάτι πρέπει να ενισχυθεί και όχι να αποδυναμωθεί. Να βρίσκουμε αυτούς τους συνομιλητές στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, να βρίσκουμε παραδείγματα και τόπους και χώρους και μέρη συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και συνομιλητέ στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσει, στα πανεπιστήμια και πρέπει αυτά να συνεχίσουμε να τα ε, καλλιεργούμε. Και εκεί μπαίνετε εσείς σε αυτό να δουλέψετε, να διατηρήσετε ανοιχτού του διάβλους επικοινωνία σε όλα αυτά τα επίπεδα. Στρέφομαι στην βουλευτή από τη Βρετάνη για να σα πω στα γαλλικά ότι ε, πρέπει να πείτε στου ε, συμπολίτε σα ότι εμεί έχουμε υπερασπιστεί τις ε, ονομασίες προέλευση. Ο, ο συνάδελφος Φιλ Χόγκαν μετά από τόσα χρόνια υπέγραψε κάτι αντίστοιχο με την Κίνα προλίγου, προλίγων ωρών και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προστατευτούν διάφορα προϊόντα ευρωπαϊκή γεωγραφικής προέλευση. Μπορείτε να πείτε στου συμπολίτε σα ότι ανοίγουμε αγορέ, όχι μόνο για τους γεωργού, αλλά και για τους υπόλοιπους, ότι υπερασπιζόμαστε την πολυμερή προσέγγιση, ότι προσπαθούμε να το κάνουμε με ανοιχτό τρόπο, με συμπεριληπτικό τρόπο, υπερασπιζόμενοι τις αξίες μας. Μπορείτε να τους πείτε ότι οθετήσαμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίσουμε και με τη δική σας βοήθεια θα συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε το δίκαιο εμπόριο σε ένα περιβάλλον κατά το οποίο οι άλλες χώρες θα δέχονται τους κανόνες, τα πρότυπα και αν δεν το πράττουν θα υπάρχουν εργαλεία για να αναγκάσουμε τις χώρες αυτές να το πράξουν. Και η κυρία Ούρσουλα Φοντεν Λάιεν, η πρόεδρος της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμεύτηκε να ε, το κάνει και να το προωθήσει. Με τη δική σας βοήθεια. Πρόκειται για μια πολιτική που βασίζεται στην εμπιστοσύνη του πολίτη. Οι τελευταίες σφίγμομετρήσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στο Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό γίγνεσθε έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ευρώπη. Αλλά δεν πρέπει να τεμπελιάσουμε, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε έτσι περαιτέρω. Τώρα, την εναλλακτική για αυτό το σώμα ε, ε, ε, εξετάσεις προσφυγών. Δεν είναι ιδανική λύση, είναι προσωρινή. Δεν βιάζονται ούτε οι άλλες χώρες να το ολοκληρώσουν αυτό και να το κάνουν. Πολλές χώρες το σκέφτονται όμως. Κάποιες χώρες περιμένουν μέχρι και την τελευταία στιγμή για να δουν. Το Δεκέμβριο θα σταματήσει να λειτουργεί το σώμα επίλυσης προσφυγών. Εάν όχι, αυτό είναι καλό. Εάν ναι, τότε θα υπάρξει επίγουσα κινητοποίηση των χωρών να δημιουργηθεί μια παράλληλη δομή που θα λειτουργεί παράλληλα και προσωρινά μέχρι ότου προχωρήσουν οι συζητήσεις με τι ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Καλά τα πράγματα με τον Καναδά και την Νορβηγία, αλλά πολύ λίγα είναι τα εμπορικά διακυβεύματα και οι εμπορικές τις επίλυτε διαφορέ με αυτέ τι δύο χώρε. Πρέπει να το διευρύνουμε αυτό. Τώρα, ε, για την πολιτική ατζέντα. Βεβαίω, η εφορία πρέπει να είναι στην πολιτική ατζέντα του ΠΟΕ με πολύ πιο συστηματικό τρόπο. Το πώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Είχαμε τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, η οποία έχει θαυτεί, πράγματι, αλλά δεν θα είναι θαμένη για πάντα. Είναι ένας τρόπος αυτός να την αναβιώσουμε για να φτιάξουμε πολιτική ατζέντα. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες χώρες στις διμερείς ή περιφερειακές εμπορικές τους συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν κεφάλαια για την αηφορία και την περιβαλλοντική αηφορία, όμως θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες αηφορίας για να μπορέσει να επιβιώσει ο ΠΟΕ. Έχω παραστεί σε διάφορα σεμινάρια, σε διάφορες επικοινωνιακές ασκήσεις, σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το πράξουμε αυτό χωρίς να μας κατηγορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες ότι βάζουμε νέους προ... κανόνες προστατευτισμού. Συνεχώς αυτό μας κατηγορούν. Ε, πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, μια δύσκολη άσκηση την οποία κάνουμε. Τώρα, εάν είπαμε την Κίνα φτάσουν σε συμφωνία. Κατά πόσο η ΕΠΑ θα θεωρηθεί ότι δεσμεύεται περισσότερο να λειτουργεί εντό του πλαισίου του ΠΟΕ. Δεν ξέρω να απαντήσω. Αυτό που ξέρω όμω είναι ότι από Ευρωπαϊκή Πλευρά ο τρόπο να λύνουμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την Κίνα, όπω είναι οι βιομηχανικέ επιδοτήσει, η κυβερνοαπάτη, η υπερβολική παραγωγή, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν και να λυθούν εντό του ΠΟΕ. Και είναι ένα από του τομεί του οποίου σημειώνουμε πρόοδο με τις ΗΠΑ ορίζουμε και προσπαθούμε να διατυπώσουμε κανόνες που θα μπορέσουμε να προβάλλουμε και στα υπόλοιπα μέλη του ΠΟΕ και να πούμε να αυτά θέλουμε να κάνουμε και να πούμε και στους Κινέζους ότι πρέπει να συμβάλλετε γιατί η πολυμερής προσέγγιση ήταν καλή για σας. Πρέπει να αναλάβετε ηγετική θέση, να αναλάβετε βούληση, να δείξετε τη βούληση να μεταρρυθμιστείτε. Αυτό πρέπει να πούμε στους Κινέζους. Και Μπορεί να μην συμφωνήσουμε σε ένα μεγάλο ψήφισμα από κοινού στην υπουργική διάσκεψη, αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια ζητήματα εργασίας, ένα πρόγραμμα εργασιών για τις μεταρρυθμίσει. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή ελπίδα προς το παρόν εν ώψη της υπουργικής διάσκεψης. Τι άλλα έχω να πω για να σκεφτώ κατά πόσο ε, το σώμα επίλυση προσφυγών, κατά πόσο θα σταματήσει να λειτουργεί ή όχι, όλο αυτό το θέμα αν θα καθυστερήσει τη διαδικασία με τα Boeing και τα Airbus. Όχι είναι η απάντηση. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια εκπρόσωπε του Ρινιού. Είστε μεροληπτικοί στην τοποθέτησή σας γιατί όντως γνωριζόμαστε επί προσωπικού από παλιά. Όμως, πράγματι πρέπει να το πούμε, το εμπόριο δεν μπορεί να λύσει ε, τη φτώχεια όλου του κόσμου ως εκθαύματος. Μπορεί όμως να βοηθήσει, να κάνει τα πράγματα πιο διαφανή, να συνδέσει τους ανθρώπους, να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι να δημιουργησει σιγά σιγά ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Είναι πεποίθησή μας αυτή. Πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης έχουν δημιουργηθεί χάρη στις εμπορικές συμφωνίες και αυτό είναι ένας τρόπος να δείξουμε στους ε, ε, ψηφοφόρους, στους συμπολίτες σας ε, συγκεκριμένα παραδείγματα. Και θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδου αξιολογήσεις για να σταλεί αυτό το μήνυμα. Σε έναν κόσμο όπου πολλές μεγάλες οικονομίες απορρίπτουν την πολυμερή προσέγγιση και το εμπόριο με βάση τους κανόνες και αρχίζουν να έχουν εσωστρέφεια, εμείς μπορούμε να είμαστε ο φάρος της ελπίδας και της υπεράσπισης αυτού του τρόπου ζωής, παρόλο που είναι ε, πιο αφηρημένο ως έννοια ε, έχουμε ε, επιχειρήματα στη φαρέτρα μας για να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, ε, ευχαριστώ για τους διερμηνείς, γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο που μας είχατε δώσει. και μπορώ λοιπόν επισήμως τώρα να πω ότι σας αποχαιρετούμε, κυρία Σεσίλια Μάλστρομ, επισήμως σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, συγχαρητήρια. Αυτές είναι αυτό είναι ο επίσημος αποχαιρετισμός μας και ο ανεπός, ανεπίσημος θα είναι στο τρίτο όροφο για ένα περιτύφ, το οποίο θα μοιραστούμε μαζί σας. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα έχουμε την Επίτροπη, την Επίτροπο μαζί μας και θα μπορέσουμε με ανεπίσημο τρόπο να συζητήσουμε για τη συνεργασία και τα αποτελέσματα στα οποία φτάσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Ευχαριστώ και πάλι, Σεσίλια. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.